Ε, καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι από εσά δηλαδή επιζήσατε μετά την πρωινή συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε συνδυάζοντας τα θέματα 21 έως 24 που αφορά την εξέταση των σχεδίων εκθέσεων ε, του Συμβουλίου που επιτρέπει την, ε, ε, την πρόσβαση διαφόρων χωρών στη σύμβαση και δίνω το λόγο στην κυρία Χάνιμπολ που είναι η συγγήτρια. Αφορά τη σύμβαση της Χάγης στις 25, 25 Οκτωβρίου 1980 οι πολιτικές πλευρές της ε, Διεθνούς Απαγωγής Παιδιού εισήχθη και η σύμβαση εισάγει ένα σύστημα συνεργασιών ανάμεσα των κρατών με σκοπό να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Πολλές φορές το πρόβλημα προκύπτει όταν οι γονείς έχουν χωρίσει. Όταν δηλαδή οι γονείς προέρχονται από διαφορετικά κράτη, υπάρχει ο πειρασμός, τα παιδιά, οι δικαιοδοσίες να διαφωνούν. Θα έχετε δει σε πολλές περιπτώσεις ε, ε, διεθνούς απαγωγής παιδιών που αφορούν χωρισμό ή διαζύγιο. Το πρόβλημα είναι η εθνική προτίμηση των νομικών συστημάτων κάθε κράτους. Και τα δικαστήρια πολύ συχνά και στα δύο κράτη ε, κηρύσουν αυτά αρμόδια για να λύσουν το θέμα. Το, προ... το... Ο σκοπός της σύμβασης είναι να επιληθεί η κατάσταση αυτή σε διεθνές επίπεδο, θεσπίζοντας ε, ότι τα αρμόδια δικαστήρια και το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το κράτος και το δίκαιο του, της χώρας ε, παραμονής του παιδιού. Και επίσης ε, προβλέπεται η άμεση επιστροφή του παιδιού που έχει απαχθεί τώρα υπάρχει και η εξωτερική αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, όπω έχει επιβεβαίωσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τα κράτη-μέλη λοιπόν δεν δρουν μόνα τους επ' αυτού και το πρόβλημα είναι ότι η σύμβαση δεν το προβλέπει και αυτή τη στιγμή έχουμε να, σκεφτούν, να αντιμετωπίσουμε τέσσερις χώρες οι οποίες έχουν καταθέσει μέσα πρόσβαση στη σύμβαση και έχουμε τώρα... Ε, το θέμα της ε, να επιβεβαιώσουμε ότι τα ενδιαφερόμενα κράτη, ή μάλλον εμείς να επιβεβαιώσουμε και να εγκρίνουμε τις προτάσεις που έχετε ενώπιόν σας για να εξασφαλιστεί ότι θα υπάρχει αυτή η προστασία για τα συγκεκριμένα παιδιά. Και εδώ στην ημερήσια διάταξη έχουμε τις εξής χώρες. Δομινικανή Δημοκρατία, η οποία υπέβαλε τον Αύγουστο του 2004 την αίτηση πρόσβασης. Υπάρχει η, προς, η πρόταση του Συμβουλίου που εγκρίνει ε, την... Ε, του Ισημερινού της Ουκρανίας, της Αυστρίας, της Κύπρου, Το, ε, ο Ισημερινός υπέβαλε στις 22 ε, Ιανουαρίου του 1992 η Ουκρανία 2 Ιουνίου του 2006 και εδώ ζητάμε από την Αυστρία σε όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του ε, Ισημερινού για κατόπιν, ε, κατόπιν έχουμε την Ονδούρα η οποία υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 1993 και συζητούμε την απόφαση του Συμβουλίου που εγκρίνει την ε, αποδοχή από την Αυστρία και την Ρουμανία. Και τέλος έχουμε την Λευκορωσία και το Πακιστάν που υπέβαλαν τον Ιανουάριο του 1998. Ε, την Λευκορωσία και το Ουσμπεκιστάν. Και και εξουσιοδοτείται η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Ρουμανία να αποδεχτούν προ το συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι διαδικαστικό θέμα, πλην όμω πολύ σημαντικό και προτείνω εμεί ω Επιτροπή να εγκρίνουμε τι τέσσερι αυτέ εκθέσει. Ε, ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Ντυράν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, για να σας ενημερώσω σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία εισηγήτρια. Είναι σημαντική διεύρυνση της Σύμβασης της Χάγης. Οι πράσινοι ανεπιφύλακτα στηρίζουν τη θέση του Συμβουλίου για την επέκταση αυτή και θέλω να διευκρινίσω, κυρία εισηγήτρια, η οποία δεν χρειάζεται να φορέσει ακουστικά γιατί γρήγορα θα ολοκληρώσω ότι δεν θα υποβάλουμε τροπολογίες και θα, ε, θα συμφωνήσουμε τη θέση του Συμβουλίου. Ε, λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας επί όλων. Ε, είμαστε τέλεια. Ε, Ο κύριος Ράντεφ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ε, η σύμβαση της Χάγης προβλέπει ότι τα θέματα της απαγωγής παιδιών Δυστυχώς υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην διερμηνία. Άρα λοιπόν είναι λοιπόν σημαντικό πάντοτε με βάση αυτή τη σύμβαση να λαμβάνεται υπόψη και η μόνιμη διαμονή των ε, παιδιών, δηλαδή το σημείο στο οποίο διαμένουν. Επίση, ε, με την προσχώρηση τη σύμβαση ε, θεσπίζεται ένα σύστημα μέσω του οποίου επιτρέπουμε την ταχεία επιστροφή των παιδιών στου γονείς τους. Για παράδειγμα, διαπιστώσαμε πολλέ περιπτώσει πέρυσι, όπω και σε άλλα χρόνια, απαγωγή ή κατακράτηση ενό παιδιού, το οποίο επισκέπτεται τον νέο γονέα μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα όπου και τα δύο κράτη σε αυτή την περίπτωση θεωρούν πως είναι αρμόδια για την εκδίκαση μιας τέτοια ε, υπόθεσης και κάθε δικαστήριο δηλαδή εκδίδει μία απόφαση για τον γονέα εκείνο ο οποίο έχει τυπικότητα του εκάστοτε κράτου μέλου. Πράγμα που δημιουργεί προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν καλώ και εγώ το ε, ε, Κοινοβούλιο να δώσει την έγκριση προκειμένου να ε, προσχωρήσουν όλε αυτέ οι χώρε στη Σύμβαση τη Χάγη. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν θέλει να προσθέσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με ευχαριστήσω απλώς την εισηγήτρια για τις εκθέσεις της. Πράγματι, η διαδικασία αυτή ξεκίνησε μετά τη γνωμοδότηση 113 ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έχουμε 14 αποφάσεις του ε, Συμβουλίου για τα κράτη και με αυτές τις τέσσερις σκοπός είναι να καταργηθεί τελείως η μεταβλητή κατάσταση που ίσχυε και την οποία επεσήμανε και στιγμάτισε ε, το δικαστήριο με την γνωμοδότηση παριθμών 13. Έτσι θα ισχύει το ίδιο νομικό καθεστώς ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, το, ε, και τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα προσθέσω τώρα ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι στο μεσημέρι της 21ης Νοεμβρίου. Καθώς δεν έχουμε τον κύριο Ντεγκράντες μαζί μας που είναι εισηγητής για το επόμενο σημείο της σημερινής σας διάταξης, αλλά έχουμε ε, μαζί μας ε, τον ε, κύριο Βόλκον, ο οποίος είναι αρμόδιος για την έκθεση υπό το σημείο 27 της σημερινής διάταξης. Ας εξετάσουμε αυτό το σημείο πρώτα, δηλαδή εξέταση των τροποποιήσεων του πρωτοκόλου υπαριθμών 3 περί του οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Βόλκον, έχετε τον λόγο. ε, αν κάτι μαθαίνει κανείς στο κοινοβούλιο είναι η ευελιξία. Οπότε εντάξει, πολύ ωραία. Θα ήθελα να, να σας ευχαριστήσω όλους ε, για τις τροπολογίες που έχετε υποβάλει. Πολύ λίγες τροπολογίες υποβλήθηκαν ε, αυτή τη φορά, μόνο πέντε. Και αυτό συμβαίνει μερικές φορές, δηλαδή τόσο λίγες τροπολογίες και νομίζω πως μπορούν να γίνουν όλες δεκτές. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, τροπολογία υπερθμών 5 που υπέβαλε ο συνάδελφος ε, Χρυσόγονος, είχα να θέσω ένα διευκρινιστικό ερώτημα γιατί με εξέπληξε λίγο. Δεν ξέρω αν παρευρίσκεται εδώ ο κύριος Χρυσόγονος. Ε, σε κάθε περίπτωση, δύο από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρούνται από την συγκεκριμένη διάταξη σε ό,τι αφορά δηλαδή τις ε, συμπερίληψη συγκεκριμένα κατηγορία δαπανών ε, των οργανισμών ε, και θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο εάν θα μπορούσε να μας εξηγήσει λίγο καλύτερα σε τι αποσκοπεί αυτή η τροπολογία. Δεν είναι όμως εδώ στην αίθουσα από ό,τι βλέπω, οπότε να πω ότι εγώ θεωρώ πως αυτές οι δύο υπηρεσίες, αυτοί οι δύο οργανισμοί δεν θα πρέπει να διαγραφούν γιατί λαμβάνεται μία απόφαση, από αυτό, λαμβάνονται αποφάσεις από αυτούς τους οργανισμούς, υπάρχει δηλαδή ένα όργανο το οποίο ε, λαμβάνει αποφάσεις, οπότε Ε, ενδεχομένως θα ε, το διευκρινίσω λίγο αυτό το ζήτημα σε ό,τι αφορά εκείνη την τροπολογία με τον ίδιο τον ε, συντάκτη της και κατά τα άλλα δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Υπάρχουν σχόλια από τα μέλη της Επιτροπής. Όχι, τότε πω η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να σχολιάσει. The stage we are addressing the... Δεν έχουμε κάποιο σχόλια. Εξετάσαμε πάντως όλες τις τροπολογίες οι οποίες ε, προτείνονται. Έχουμε αρχίσει να σχηματίζουμε τη δική μας άποψη σε σχέση με αυτέ και όταν θα περάσουμε στο φάση του τριμερούς διαλόγου θα εκθέσουμε τις δικές μας θέσεις. Καλώς λέει ο πρόεδρο. Τώρα ο, παρευρίσκεται εδώ ο κύριο Ντεγκράντε ε, Πασκουάλ στην αίθουσα, οπότε επιστρέφουμε στο προηγούμενο σημείο τη ημέρα διάταξη, δηλαδή Σημείο 26. Εξέταση σχεδίου έκθεση σε ό,τι αφορά το συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασία για τα φάρμακα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Τεγκράντη Πασκουάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την αργοπορία. Έπρεπε να ασχοληθώ με άλλα αναπόφευκτα θέματα. Θα σας μιλήσω λοιπόν ως εισηγητής για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα ήθελα καταρχήν να σας μιλήσω για ένα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, αλλά που ε, γνωμοδοτούν και η ΕΜΒΗ και η ΙΝΤΑ. Θα σας μιλήσω για το ιστορικό της ε, υπόθεσης επίσης. Η στρατηγική της Επιτροπής για την ενιαία αγορά ε, όρισε εξαιρέσεις σε αυτό το πλαίσιο για να αυξαθεί, αυξηθεί συγγνώμη, η ανταγωνιστικότητα των ε, γενώσιμων και των βιοομοιδών φαρμάκων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εξαγωγή. Και έτσι οι αγορές της Ευρωπαϊκής, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να προωθήσουν αυτά τα γενώσιμα φάρμακα. Η απόφαση λήφθη το 2016 και προσπαθήσαμε να προτρέψουμε την Επιτροπή να εισαγάγει πριν από το 19 μία ε, εξαίρεση για να μπορούμε να προωθήσουμε την ε, ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στον τομέα της παρασκευής φαρμάκων, ιδιαίτερα γενώσιμων και ορίζοντας ένα ειδικό καθεστώς για τα βιομοειδή και τα γενώσιμα φάρμακα. Η Επιτροπή τώρα προτείνει την αλλαγή του κανονισμού του 2009 σε σχέση με την επιπλέον πιστοποίηση των φαρμάκων για αυτή την εξαίρεση παρασκευής προς εξαγωγή. Έτσι, στο μέλλον, οι επιχειρήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσουν να παρασκευάζουν ε, γενώσιμα ή βιοομοειδή φάρμακα κατά την περίοδο αυτή. Αυτό μόνο για εξαγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εισηγητής ε, θέλω να δω και θέματα πολιτικής υφής Θεωρώ δηλαδή ότι μπορούμε έτσι να άρουμε ένα πρόσκομα σε σχέση με την παρασκευή γενώσιμων φαρμάκων, έτσι ώστε να έχουμε ίση πρόσβαση στην αγορά όσο αφορά την παρασκευή αυτών των φαρμάκων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι φτάνουμε σε μια συμφιλίωση συμφερόντων που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Αυτό προσπάθησα να κάνω και στην έκθεσή μου. Να δω ποιες είναι οι επιλογές που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα του φαρμακευτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατανοώ όλες τις απόψεις, ακόμα και τις αποκλίνουσες και δεν θεωρώ ότι ότι υπάρχει διχοτόμηση μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων και των ε, φαρμακευτικών εταιριών που παρασκευάζουν γενώσιμα. Και από εκεί ορμόμενος προβάλλω αυτή την πρόταση έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελεί δέλεαρ για τις επενδύσεις και για να εγγυηθούμε την ανταγωνιστικότητα για τους παρασκευαστές γενώσιμων και βιομοιδών φαρμάκων για να μπορούν να τα εξάγουν στην παγκόσμια αγορά. Και ακριβώς αυτό καλύπτουν και οι τροπολογίες μου, έτσι ώστε να εξορθολογήσω αυτό το πλαίσιο εφαρμογής, έτσι ώστε η πρόταση να είναι αναλογική ε, και δίκαιοι καθώς και ισορροπημένη, με βάση την πρόταση της Επιτροπής. Γι' αυτό υπάρχει και ένα παράρτημα έτσι ώστε να ενημερώσουμε τους παρασκευαστές γενώσιμων για την προστασία εμπιστευτικών στοιχείων ή ευαίσθητων στοιχείων έτσι ώστε οι παρασκευαστές να έχουν τις πληροφορίες για να δουν κατά πόσο πληρούνται οι συνθήκες για την χορήγηση αυτής της εξαίρεσης και για να μην πλήτεται ο ανταγωνισμός. Για να μπορέσουν τα συμβαλόμενα μέρη να έχουν χρόνο για να επαληθεύσουν την πιστοποίηση αυτή, προτείνω να διευρύνουμε την ε, προθεσμία σε τρεις μήνες έτσι ώστε οι φαρμακοβιομηχανίες να μας ενημερώσουν για τα γενώσιμα και τα βιομοειδή. Άρα θα έχουμε το κείμενο έτσι ώστε να ξέρουμε ότι η αρμόδια αρχή πιστοποίησης και έβρεση τεχνίας μπορεί να μας δώσει όλα τα στοιχεία που προαπαιτούνται. Επίσης θα υπάρχει και ε, ένα νέο δελτίο, μία νέα φόρμα που θα πρέπει να συμπληρώνεται και έτσι έχουμε και το παράρτημα ένα της πρότασης σε σχέση με τις πληροφορίες του παρασκευαστή. Λαμβάνουμε υπόψη την υποχρέωσή του να ενημερώσει τους υπεύθυνους των βιομοιδών ότι πρόκειται για ε, πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Σε σχέση τώρα με την θέση σε ισχύ, η εξαίρεση ισχύει για τη, τις πιστοποιήσεις των οποίων το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λύγει μετά το 2023 για να μην υπάρχει νομικό χάσμα και να υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο που να ισχύει για την εξαίρεση. Επίσης υπάρχει μεγάλη μεταβατική περίοδος έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες επενδύσεις και οι φορείς της αγοράς να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες της αγοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Λοτόφσκι. Ε, ε, δύο λόγια εκ μέρους του ECR. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεγκράντες Πασχουάλ για την σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης. Δεν βλέπουμε να υπάρχει μεγάλη διαφορά στις θέσεις που παρουσιάστηκαν και στις θέσεις της ομάδας μας. Θα χρησιμοποιείτε ένα ενιαίο έντυπο. Και πρέπει να ξεκαθαρίζονται κάποιοι ορισμοί που βεβαίως ε, εξορθολογίζουν τις διατάξεις συνεργασίας μεταξύ πολλών αρχών. Συμφωνούμε ότι αυτή η γνωμοδότηση ή μάλλον αυτή η έκθεση αφορά τη δυνατότητα να αυξηθεί ο όγκος παραγωγής των γενοσύμων στην Ένωση και να τους επιτρέπει να γίνουν ανταγωνιστικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντιλαμβανόμαστε ότι δύο είναι οι κατηγορίες των εταιριών. Αυτές που παρασκευάζουν τα γενώσιμα και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Επίσης, θέλουμε να συζητήσουμε και την, την καταληκτική ημερομηνία που παρουσιάστηκε, αλλά και την ε, καταληκτική ημερομηνία για την εφαρμογή των διατάξεων. Φυσικά θα υποβάλουμε τροπολογίες, όμως δεν διαπιστώνουμε να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην έκθεση του εισηγητή. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την πρόταση με την αλλαγή αυτού, του, αυτής της νομοθεσίας σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό προστασίας για τα φάρμακα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ίσους όρους του παιχνιδιού, αν θέλετε, για τους, ε, ε για τους ε, παρασκευαστές, δηλαδή φαρμάκων, ειδικότερα ε, γενοσύμων και βιομοειδών ε, και εντό και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο χαιρετίζουμε ιδιαίτερα ως στόχο σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, τις οποίες δεν υπάρχει ε, μια προστασία αυτού του είδους, του συμπληρωματικού δηλαδή πιστοποιητικού ε, ε, προστασίας, κάνουμε ακριβώς τη σωστή κίνηση και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό γενικότερα το ζήτημα των ε, φαρμάκων, το οποίο έχουμε υπογραμμίσει και πάλι ε, με την μορφή δύο νομοθετήσεων από την πλευρά, ε, συγγνώμη, δύο ψηφισμάτων, ψηφισμάτων από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δείχνουμε να δίνουμε συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Ωστόσο, θεωρώ πως λείπει μια σημαντική πτυχή από αυτή την έκθεση. Αναφέρεται δηλαδή Αναφέρονται δηλαδή ε, όλα αυτά ε, που αναφέρονται μέσα στην έκθεση, αλλά όχι το γεγονό ότι είναι πολύ θετικό για του ίδιου τη πολίτε τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την περίπτωση του stockpiling, τη αποθήκευση. Δηλαδή, θα πρέπει να προβλέψουμε αντίστοιχη ρύθμιση όχι μόνο για τι εξαγωγέ, αλλά και για το stockpiling. Και αυτό για να σεβαστούμε και τα ίδια τα ψηφίσματα που εμείς από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουμε εμ, υιοθετήσει. Επίσης θεωρούμε πως ε, ε, από εκεί και μετά η πρόταση του να καταστούν πιο αυστηρές οι υποχρεώσεις ε, ε υποβολής εκθέσεων είναι κάτι το εσφαλμένο και θα υποβάλουμε και τροπολογίες ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι η έκθεση και η πρόταση έτσι όπως θα πρέπει να γίνει θα πρέπει ακριβώς να κατευθυνθεί λίγο περισσότερο προς το όφελος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιλαμβάνομαι ότι βέβαια είναι αμφιλεγόμενη αυτή η πρόταση ε, που προετοιμάζουμε ε, τώρα ε, στην φαρμακοβιομηχανία. Δηλαδή, από τη μία πλευρά έχουμε εκείνου που παρασκευάζουν γενώσιμα και από την άλλη πλευρά του originators, δηλαδή εκείνου που κατασκευάζουν τα πρωτότυπα φάρμακα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σε οποιαδήποτε πρόταση, θα πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου και του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια σε αυτή την πρόταση, κατά τη δική μα άποψη, θα πρέπει να περιληφθεί και η αποθήκευση, το stockpiling. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Η Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εμείς θέλουμε καταρχήν να πούμε ότι είναι ευπρόσδεκτη η, το σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει πολλές διευκρινήσεις, συγκεκριμενοποιήσεις ε, και άλλα πολύ χρήσιμα που θα βελτιώσουν την πρότασή μας. Θα ήθελα να πω με δύο λόγια κάποια θέματα που μας προκαλούν ανησυχία ή ερωτήματα, αν θέλετε. Στην πρόταση υπάρχει τροπολογία που λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμό για τι εμπιστευτικέ πληροφορίε. Πράγματι θεωρούμε το στόχο σοβαρό. Αν δείτε το καθεστώ κοινοποίηση, θα ήταν καλύτερα να προσδιοριστεί στο πλαίσιο του καθεστώτο αυτού Πώ θα αντιμετωπιστεί το θέμα για μα, Αυτό θα πρέπει να μεταφραστεί ω εξή. Ποιο θα παίρνει ποιε πληροφορίε, πότε κλπ. Και να μην υπάρχει μια γενική διάταξη που θα λέει ότι δεν μπορεί να διαβιβάζονται εμπιστευτικέ πληροφορίε. Αυτό από μόνο του θα οδηγήσει σε νομική αβεβαιότητα. Ο στόχος είναι θετικός, αλλά πιστεύω, πιστεύουμε ότι πρέπει να διατυπωθεί ε, διαφορετικά και να ενταχθεί στο, στο κείμενο της πρότασης. μια δεύτερη μικρότερη ανησυχία, αλλά μιλάμε τώρα για λεπτομέρειες και γι' αυτό δεν θέλω να σας καθυστερήσω και πολύ. Ο κατάλογος των τρίτων χωρών. Στη δική μας πρόταση ο κατάλογος τρίτων χωρών πρέπει να ε, δημοσιεύεται, όμως δεν είχαμε στην πρότασή μας την υποχρέωση να διαβιβάζεται ο κατάλογος αυτός με τον κάτοχο του πιστοποιητικού. Εδώ η συγητής το αντιέστρεψε εντελώς και μας δημιουργεί μια ανησυχία το ότι αυτές οι πληροφορίες θα πηγαίνουν στον ουσιαστικά ανταγωνιστή του κλάδου ακριβώς για τους λόγους που επεσήμανε στην έκθεση και ο εισηγητής. Αυτό μπορεί να αποτελεί ε, εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. Έτσι λοιπόν φτάνει σε έναν εμπορικό εταίρο χωρίς να έχουν δημοσιευτεί. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η βάση προσέγγισης. Μπορεί να είναι προβληματικό στον τομέα του ανταγωνισμού. Και τέλος, αν μου επιτρέπετε, σχετικά με το χρόνο, ε, σημειώνουμε το ενδιαφέρον για την, τις πρότασεις και τις προτάσεις του εισηγητή. Θα θέλαμε όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια λεπτή ισορροπία. Ανάμεσα αφενός σε αυτόν που ενδεχομένως είναι επιθυμητό από οικονομική και πολιτική σκοπιά, αλλά και από ότι είναι ε, εφικτό νομικά, γιατί έχουν χορηγηθεί δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν να προστατευτούν οι δικαιολογημένες προσδοκίες. Και αν θέλουμε να εισάγουμε μια εξαίρεση, αυτό πρέπει να δικαιολογείται προσεκτικά υπό το φως των ε, λόγων δημοσίου συμφέροντος. Έτσι λοιπόν, αν θέλει το Κοινοβούλιο να μπει σε αυτή την προσπάθεια, θα πρέπει να είναι απολύτως σαφές. Και με τις μικρές αυτές επιφυλάξεις θα ήθελα να πω ότι για μας είναι ευπρόσδεκτη η ε, δουλειά αυτή και θα συζητηθεί, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμπληρώσω τις πληροφορίες λέγοντας ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 23η ε, Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα. Οπότε, κύριε Ντεγκράντες, θέλετε τον λόγο? Ναι, εντάχει, πρόεδρε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εκτιμώ την αξία των παρεμβάσεων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του ECR ως προς τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές ε, σημείωσα αυτά που είπε ως προς τη διασάφηση ισχύ του κανονισμού καθώς και τα στοιχεία αποφασιστικής σημασίας για να φτάσουμε σε μία εξισορρόπηση ως προς την επαόριστο αναβολή, την αναβολή συνεντίε και στην περίπτωση αυτή θα το δούμε μεταξύ Νομίζω ότι και οι σοσιαλιστές έκαναν μία πολύ ισορροπημένη παρέμβαση. Αλλά εδώ ε, έχουμε να κάνουμε με τη διαφορά μεταξύ καινοτόμων και γενώσιμων ε, φαρμάκων που αποθηκεύονται. Αυτό είναι και θέμα ονοματολογίας, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ε, ονοματολογία τάσεται υπέρ των γενώσιμων. Είχαμε αυτή την προθεσμία πέντε ετών μετά τη λήξη του διπλώματος Τεχνίας και αυτό ήταν υπέρ των καινοτόμων διότι εν οι παρασκευαστές των ε, καινοτόμων φαρμάκων πρέπει να έχουν μία κάλυψη τη στιγμή που έχουν δίπλωμα Τεχνίας. Τώρα όμως, με στα πλαίσια της πενταετίας, τι κάνουμε. Ε, καλύπτουμε την συμμετοχή των ε, γενώσιμων. Δηλαδή υπάρχει ένας λόγος μεταξύ καινοτόμων και γενώσιμων για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν τους παρασκευαστές τρίτων χωρών. Το ίδιο αφορά και την Παρασκευή και την αποθήκευση. Τώρα, τι γίνεται με την αποθήκευση. Εδώ δεν πρέπει να υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Βρίσκεται πέρα από την ισορροπία στην οποία έφτασε η Κομισιόν. Το θέμα της αποθήκευσης. Εγώ θεωρώ ότι η πρόταση της Επιτροπής ήρθε αργά, γιατί είναι πολυσχηδές το ζήτημα και μας παρουσιάζει την ε, πρόταση σε ένα κάκιστο χρονικό διάστημα, σε μία κακή πολιτική συγκυρία τη στιγμή που υπάρχει συναπόφαση και πρέπει να φτάσουμε σε συνδυασμού. χωρίς να υπάρχει διασταλτική ερμηνεία. Όμως οι πολιτικές ομάδες ξέρουν ότι αυτό είναι μία ανάγκη για την Ευρώπη για να είναι ανταγωνιστική με τον υπόλοιπο κόσμο και να μην υπάρχουν τόσα προσκόμματα. Καταγράφω αυτά που θέλετε να συζητήσουμε. Αυτό το λέω προς τους ε, σοσιαλιστές αλλά θα δούμε και θα αποτιμήσουμε όλα τα στοιχεία παρασκευής και αποθήκευσης. Ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μία υφέρπουσα επιφυλακτικότητα. Υπάρχει το νούμερο κλάουσους ή είναι ανοιχτός ο αριθμός συμμετοχών. Αυτό θα πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Φαίνεται ότι η Επιτροπή είναι επιφυλακτική αυτή τη στιγμή. Δεν πρέπει να εισραίουν υπερβολικά πολλά στοιχεία που να αποτελούν πρόσκομα στον ανταγωνισμό. Αλλά υπάρχει και το θέμα της νομικής ασφάλειας. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε πλήρη στοιχεία, τότε μπορεί να ανακύψουν διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Κάτι το οποίο πρέπει να αποφευχθεί. Θα το δούμε με τους σκιώδεις, και θα ε, εξετάσουμε τις τροπολογίες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα φτάσουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες. Μέσα στα πλαίσια αυτού του ε, ε, ιδιαίτερα αρνητικού χρονισμού μέχρι τον Απρίλιο για την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και τον νόμιμο συμφέρον των παρασκευών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Μέσα στο πλαίσιο της, ελευθερίας, ε, της ευελιξίας που ανέφερε ο κύριος Βέλκεν και επειδή λείπουν δύο εισηγητές ε, που, των δύο επόμενων θεμάτων, θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, για το θέμα 30 που αφορά τη μελέτη των ε, τροπολογιών για τις αντιπροσωπευτικές δράσεις για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων στον κύριο Δίγκη. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάζω με συνενοχή τη Μαρή Ντελβό, τη δεύτερη, στη δεύτερη συνάντηση των σκιωδών πριν από λίγα λεφτά μπορώ να πω, αλλά αυτό με δική μου, δική μου αισιοδοξία, ότι κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση, είμαστε σε καλό δρόμο και ότι ελπίζω μετά τη συνεδρίαση αυτή θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία με για ένα καλό ισορροπημένο κείμενο που θα προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την ασφάλεια των επιχειρήσεων. Δεν πρέπει να κάνουμε το ένα χωρίς το άλλο. Στα σημεία συμφωνίας τα οποία ε, βρέθηκαν, ένα αφορά την ελάχιστη εναρμόνιση. Δεν θέλω να επιβάλλω δηλαδή στα άλλα κράτη-μέλη κανόνες ασυμβίβαστους με τα, με τα συνταγματικές τους διατάξεις και γι' αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό το δικαίωμα της διαδικαστικής αυτονομίας που έχουν τα κράτη-μέλη. Άρα είναι η αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης. Το δεύτερο σημείο συμφωνίας είναι η παροχή εξαίρεσης σε κάποιους οντότητες για να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένα νομικά συστήματα. Ο Ombudsman των κάποιων βορείων χωρών, όπως η Δανία, όπου πρέπει να παίξουν το ρόλο του αρμόδιου οργανισμού εκπροσωπώντας ε, τον συγκεκριμένο οργανισμό που αναφέρουμε στο σχέδιο. Τρίτο, τρίτη περίπτωση συμφωνίας εκ πρώτης όψεως, παρότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν ε, διευθετηθεί είναι η δημιουργία των διατάξεων που θα διαφυλάξουν την εργαλειοποίηση οποιασδήποτε αντιπροσωπευτικής δράσης. Άρα ε, καθορίζουμε και εξελίσσουμε κριτήρια διαφάνειας όσον αφορά τη ε, χρηματοδότηση και τα σύγκρουση συμφερόντων για τους αρμόδιους οργανισμούς. Επίσης, άλλο σημείο συμφωνίας. Προχωρούμε προς μια κοινή αντίληψη για μια ισορροπία που θα κάνει ε, περιοριστικούς τους όρους της φιλικής διευθέτησης και ταυτόχρονα ελήψη αυτού να υπάρξει ατομική προσφυγή. Τέλος, last but not least, λέει ο μιλήτης, συμφωνούμε ε, επί της αρχής του loser pays, δηλαδή αυτός που χάνει πληρώνει, γιατί είναι σαφές ο καθένας να αντιμετωπίζει τις ευθύνες του. Ε, φυσικά μένουν ακόμα πράγματα να γίνουν. Υπάρχει καλή θέληση από όλες τις πολιτικές ομάδες και ευχαριστώ ειλικρινά και του ε, της, τους σκιώδης εισηγητές, είπα για τη Μάντι, αλλά και τις όλες τις ομάδες και οι συνάδελφοι βουλευτές, τα μέλη, αλλά, αλλά και όλοι όσοι δουλεύουν γνωρίζοντας απόλυτος το θέμα τους και φροντίζουν τις λεπτομέρειες και φροντίζουν ε, να σέβονται τις κόκκινες γραμμές των πολιτικών ομάδων και να βρίσκουν μια συμφωνία που θα οδηγήσει σε πλειοψηφία. Μίλησα τις, ε, για τις κόκκινες γραμμές των πολιτικών ομάδων. Η δική μου πολιτική ομάδα έχει ως κόκκινη γραμμή την αρχή του opt-in. Όμως και πάλι θα προσπαθήσουμε να, βρεθούν, να βρεθεί ισορροπία ώστε να προχωρήσουμε με βάση τη λογική και προς την καλύτερη κατεύθυνση που είναι η προστασία του καταναλωτή. Στόχος μας είναι να ολοκληρωθεί το κείμενο ως το δυνατόν ταχύτερα, ώστε αυτή η μεταρρύθμιση που για, για μένα είναι από αποφασιστική σημασία στην προστασία των καταναλωτών να βοηθήσει να γίνει πιο προστατευτική η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ κυρία Ντοβού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, διαπιστώσατε ότι υπάρχει αρμονία ανάμεσα στον κύριο Τιτιέ και ε, σε μένα. Θέλω να επισημάνω ότι πράγματι έγιναν δύο συναντήσεις και μέχρι στιγμής προχωρούμε καλά. Όπως όλοι γνωρίζουμε όμως, τίποτα δεν έχει τελειώσει αν δεν έχουν όλα ε, διευκρινιστεί. Εν πάση περιπτώσει, θέλω και όπως και εκείνος να ευχαριστήσω τις ομάδες αυτών που εργάζονται για το, επί του θέματος Πράγματι, τρία θέματα εγώ θέλω να θίξω. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε ο εισηγητής, όμως όλοι έχουμε τον ίδιο σκοπό, να βρεθεί μια ισορροπία, αφενός ώστε οι εκπρόσωποι να έχουν την δυνατότητα να αναλαμβάνουν δράση ως αντιπρόσωποι, αλλά και να εξασφαλίσουμε κάποιες εγγυήσεις της επιχειρήσεις. Αυτό είναι το common ground, ο κοινό τόπο επί του οποίου δουλεύουμε. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για ισορροπία και να μην καταστούν αδύνατες οι αντιπροσωπευτικές δράσεις, γιατί στόχος είναι η προστασία του καταναλωτή να έχει μέσα δράσεις αυτό που με ενοχλεί εξ αρχής είναι ότι κάποιες τροπολογίες δείχνουν ότι εκ των προτέρων ε, υποψιάζονται ότι θα υπάρξει χειραγώγηση από επικίνδυνους καπιταλιστές, ανταγωνιστές κλπ. Έτσι διαβάζω κάποιες τροπολογίες. Δεν είναι αυτό το πνεύμα ε, με το οποίο θα πρέπει να ε, συνταχθεί αυτή η οδηγία. Φυσικά δεν αναφέρουμε στον κύριο Ντιντιέ, δεν λέω ότι αυτή είναι τη του, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να βρεθεί η ισορροπία, σωστή ισορροπία. Το δεύτερο θέμα είναι ότι χαιρετίζω το συμβιβασμό που προτείνει ο εισηγητής να προταθεί ε, μια ελάχιστη, να έχει ένα ελάχιστο χαρακτήρα αυτό που προτείνει η οδηγία, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε καλύτερα και να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες ε, στην υπεράσπιση των καταναλωτών με το ίδιο πνεύμα είναι ευπρόσδεκτη η, η πλευρά της επικουρικότητας που περιλαμβάνει η οδηγία και που μας προσφέρει η Κομισιόν. Και για τον λόγο αυτό δεν είμαι υπέρ του να υποχρεωθούν τα κρατη να ε, επιλέξουν είτε opt-in είτε opt-out. Γιατί εξ όσων γνωρίζουμε υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα στα κρατη Και δεν νομίζω ότι μια οδηγία που σκοπό έχει την προστασία των καταναλωτών θα, θα έπρεπε να επιβάλλει σε ένα κράτο μέλος να αλλάξει την παράδοσή του και να αλλάξει μια παράδοση για να χρησιμοποιήσει ένα opt-in ή ένα opt-out. Η μόνη εναλλακτική που θα ήθελα να επιτρέψω είναι ο καταναλωτής άλλου κράτους μέλους να μπορεί να κάνει opt-in αν το επιθυμεί και να ενταχθεί σε μία αντιπροσωπευτική δράση ε, ενός κράτους μέλους το οποίο δεν ε, κατοικεί. Ας πούμε, ας πούμε ότι κατοικεί σε μια χώρα, αλλά αν θέλω να ενταχθώ σε μια class action, σε μια αντιπροσωπευτική δράση της στη Γερμανία, θα μπορώ να το κάνω και βεβαίως εκεί υπάρχει το opt-in. Το τρίτο σημείο και τελευταίο, Θέλω να υπενθυμίσω ότι η ομάδα μου θέλει να διευρύνει το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία και όχι να το περιορίζει μόνο στους καταναλωτές. Για ποιο λόγο, για ποιο λόγο διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή, επειδή θέλαμε, επιθυμούμε να εισάγουμε την ε, περιβαλλοντική βλάβη και την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Στις ε, περιπτώσεις αυτές τα θύματα δεν είναι όλοι καταναλωτές. Υπάρχουν πολλοί που εμπλέκονται, στους οποίους αφορά και θα ήθελα πολύ να μπορέσουμε ε, να κάνουμε αυτή την προσθήκη στο κείμενο. Κατόπιν αυτού είμαι αρκετά αισιόδοξη ότι θα καταλήξουμε σε εύθετο χρόνο σε ικανοποιητική συμφωνία. <laughs> Ευχαριστώ. Thank you as well, uh, Monsieur Le Breton. Ευχαριστώ, κύριος Le Breton. Oui, tout d'abord, je veux dire qu'il m'est θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ ευχάριστο να συμμετέχω σε μια συζήτηση όπου επικρατεί η γαλλική γλώσσα και δεν χρειάζεται να βάζω ακουστικά. Ευχαριστούμε κύριε Ντιντιέ για αυτή την παρουσίαση. Ε, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο γιατί αναγνωρίζω αυτά που είπατε ως ε, προς την διαδικαστική αυτονομία των κρατών μελών. Αυτό είναι πολύ θετικό, δέχομαι αυτή την προσέγγιση. Υπάρχουν όμως και ορισμένες συνέπειες που διαφέρουν από τις δικές σας. Αφήνουμε σε κάθε κράτος την επιλογή του opt-in ή out ανάλογα με την παράδοσή του. Όπως είπε και η κυρία Ντελβό, αν επιβάλλουμε μια λύση ε, σε, στα κράτη, δεν τηρούμε την ελάχιστη εναρμόνιση. Ε, θα ήθελα, και ίσως να μην το δέχεται η κυρία Ντελβό αυτό, θα ήθελα να ασχοληθούμε με την προστασία των καταναλωτών, αλλά όχι υπό τη στενή έννοια ε, σε σχέση με το περιβάλλον ή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Νομίζω ότι προτρέχουμε ε, δεν θα πρέπει να είμαστε υπέρμετρα φιλόδοξοι. Βρισκόμαστε στο τέλος της θητείας και αν θέλουμε να συμφωνήσουμε επί ενός κειμένου θα πρέπει να ε, οριοθετήσουμε το θέμα μας και να μην κάνουμε παρεκβάσεις. Ε, η κυρία Ντελβό υπορισμένα πράγματα που δεν με βρίσκουν σύμφωνος. Νομίζω ότι στις συλλογικές προσφυγές υπάρχει και ένα στοιχείο χειραγώγησης και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όπως είπε και ο κύριος Διδιέ θα πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε παράλογοι. Άρα Συμφωνώ και με αυτή την προληπτική αρχή. Η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ανοίγουμε ε, ένα μεγάλο ε, δρόμο για την ε, προσφυγή στα, στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ε, κατοίκων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μη κατοίκων. Και αυτό προέκυψε από το μεγάλο σκάνδαλο της Volkswagen. Υπάρχουν συλλογικές προσφυγές και ένδικα μέσα σε πολλά κράτη υπέρ των καταναλωτών. Θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Δεν συμφωνούμε πάντα όλοι, αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτή η πτυχή του θέματος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επικοδομητική προσέγγιση ως προς τις προγενέστερες, προγενέστερες συζητήσεις. Είναι αχαρτογράφητα αυτά τα ύδατα, γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας καινούργιας πραγματικότητας. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας ε, για να μην υπάρχει κατάχρηση του μηχανισμού. Σημεριζόμαστε αυτές τις ανησυχίες. Από την άλλη πλευρά ε, υπάρχουν καταχρήσεις ως προς τις συλλογικές ε, προσφυγές. Ε, το Οργανισμός Προστασίας των Καταναλωτών όμως στην Ευρώπη δεν μπορούσε να μου δώσει παραδείγματα αυτής της κατάχρησης. Εάν υπάρχουν να μου το πείτε. Υπάρχουν ε, βεβαίως και μεγάλες επιτυχίες σε περίπτωση υπερβάσεων ή ε, εγκληματικών δράσεων. η αρχή του ότι ο, ο φιλέτης, αυτός που χάνει, καταβάλει το τίμημα, το αντίτιμο, θα πρέπει να φτάσουμε σε μία λύση όπου ο εθνικός δικαστής θα αποφανθεί. Άρα θα πρέπει να υπάρχει υπενθύμηση προς όλους που χρησιμοποιούν αυτό το μέσο της ε, συλλογικής προσφυγής ότι ε, θα πρέπει να χύσουν δάκρυα, υδρότα και αίμα. Και σε πολλές περιπτώσεις διανοίγεται μία νέα οδός για καλύτερη νομοθέτηση και δικαιοσύνη. Άρα θα πρέπει να γίνει εξισορρόπηση και εδώ. Δεν θα πρέπει να προσπαθεί προσπαθήσουμε να ε, οδηγήσουμε σε μία αποδόμηση της λειτουργίας στα κράτη-μέλη. Ίσως θα μπορούσαμε να δούμε και ορισμένες χριστές πρακτικές από τα κράτη-μέλη και να τις εντάξουμε σε αυτό το μηχανισμό. Βλέπω πρόοδο στις διαπραγματεύσεις και νομίζω ότι στο εγγύς μέλλον θα υποβάλουμε μια πολύ καλή πρόταση. Ο κύριος Διντιέ παίρνει πολύ σοβαρά το ρόλο του, ο κύριος Βος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τον εισηγητή. Πράγματι μπορώ να τα επιβεβαιώσω αυτό που αναφέρθηκε σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και την προσέγγιση που ακολουθείτε και την οποία θεωρώ πολύ θετική, δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνει ένας διάλογος με όλους. Παρ' όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι σε ό,τι αφορά την πρόταση που γίνεται εδώ, σε ό,τι αφορά τη συλλογική προστασία, δεν επιλύονται δύο βασικά προβλήματα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το νέο σύστημα των αντιπροσωπευτικών δρόσεων θα υπάρχει συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα αλλά σε νοσιακό επίπεδο με πολύ λιγότερες, πολύ πιο περιορισμένες προστατευτικές διατάξεις. Σε σύγκριση δηλαδή με ό,τι προβλέπεται σε εθνικό επίπεδο. Άρα κανείς δεν θα προτιμάει μια τέτοια ενωσιακή δράση και κατά συνέπεια εκ των πραγμάτων η προτίμηση θα είναι πάντοτε υπέρ των εθνικών ε, δράσεων. Οπότε θα πρέπει λίγο να προσέξουμε καλύτερα πώς θα προβλέψουμε ε, κάτι τέτοιο. Ε, δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Επιτροπή με την πρότασή της ε, διευκολύνει πλέον ε, την υποβολή ε, τέτοιου είδους δράσεων από την πλευρά κερδοσκοπικών φορέων, οι οποίοι δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για το συμφέρον των καταναλωτών, αλλά ακριβώς για το δικό τους κέρδος. Και αυτό το πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε τη σήμερα ημέρα στις κάτω χώρες, όπου δηλαδή βλέπουμε ακριβώς να υπάρχει αυτό το ελεύθερο πεδίο και να εμφανίζονται τέτοιου είδους φορείς κερδοσκοπικοί, οπότε ε, δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε ένα τέτοιο σφάλμα σε νοσιακό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτού τους κινδύνου που θα μπορούσαν να προκύψουν με βάση την πρόταση τη Επιτροπή. Κατά τη δική μου άποψη, για να του αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να ε, καταστούν πολύ πιο αυστηρές οι δικλείδες αυσαλία τη ε, πρόταση τη και να είναι πιο περιορισμένο το πεδίο. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να υπάρχει και καλύτερη ρύθμιση τη ε, Συνεργασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ των εθνικών συστημάτων δράσεων και του ενωσιακού. Ε, θα πρέπει να προβλέψουμε διατάξεις, για παράδειγμα, οι οποίες θα αποκλείουν το forum shopping, δηλαδή το να επιλέγει κανείς ε, που μπορεί να δραστηριοποιηθεί και αυτό μπορεί να γίνει με τροποποιήσει στα άρθρα 1, 2, 6 και 16, ειδικότερα στο ένα που αφορά το πεδίο εφαρμογή και στο παράρτημα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να περιορίσουμε κάπω και του σχετικού ορισμού που έχουμε. Σε ό,τι αφορά το, τη σχέση τώρα ανάμεσα στο ενωσιακό σύστημα και τα εφιστάμενα εθνικά συστήματα, θα πρέπει αυτή να διευκρινίζεται ε, πλήρω και να μην δίνονται δυνατότητε παράλληλη. Ε, σε τέτοιων δράσεων. Και σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές περιπτώσεις θα πρέπει να ορίζεται και η δικαιοδοσία του αρμοδίου δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 4 και τα qualified entities, θεωρώ πως θεωρούμε εδώ πως είναι απαραίτητα πολύ αυστηρά κριτήρια ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το ιστορικό και την διάρθρωση ενός τέτοιου φορέα, ε, ούτω ώστε να καταδεικνύει ότι πράγματι ο εν λόγω φορέας ε, έχει ένα νόμιμο συμφέρον σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών και επίση θα πρέπει να έχουν αυτόνομο χαρακτήρα και να μην συνδέεται είτε δομικά είτε μέσω σύμβασης με άλλους φορείς, για παράδειγμα οικονομικής φύσης ή επενδυτικής φύσης και βέβαια σε επίπεδο ε, και οργάνωση και σε επίπεδο προσωπικό θα πρέπει να διαθέσετε την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη. Σε ό,τι αφορά τώρα το άρθρο 6 και την δυνατότητα του opt-in σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές ε, αντιπροσωπευτικές δράσεις, ε, θεωρώ πως εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο αριθμός συμμετεχόντους ώστε ακριβώς να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την διαφοροποίηση ανάμεσα στα εθνικά συστήματα και το ενωσιακό επίπεδο για να γνωρίζει κανείς επάντοτε πότε μπορεί να κινηθεί σε εθνικό επίπεδο και πότε σε ενωσιακό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αν θα πρέπει να ε, δραστηριοποιηθεί και ε, στις δύο δράσεις ε, και θα υπάρχει κατασπαστάληση των, των, των σχετικών κονδυλίων, αλλά και θα υπάρχει περισσότερο διοικητικό άχθος. Άρα λοιπόν οι τροπολογίες που εγώ υποβάλλω κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και επίσης ένα ακόμα άρθρο που μας απασχολεί είναι το άρθρο 7 σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της διαδικασίας. Θεωρούμε πως ε, αυτή η διαδικασία θα πρέπει να είναι απαγορευμένη για εμπορικού χαρακτήρα επενδυτές. Δηλαδή δεν θα πρέπει να είναι δυνατό να αντλήσει κανείς σε κέρδος από μια τέτοια συλλογική δρασιαγωγή. Προφανώ οι δικηγόροι θα πρέπει να αμείβονται και υπάρχουν σχετικέ διατάξει, αλλά το ποσό, για παράδειγμα, το οποίο μπορεί κανεί να κερδίσει μέσω μια αγωγή, θα πρέπει να προορίζεται για του ίδιους τους καταναλωτέ και όχι ω κέρδο. Και γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, Ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί έτσι ώστε να μην προβλέψουμε ένα σύστημα το οποίο στην πράξη δεν θα οδηγήσει σε υψηλότερη προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Από πλευράς Επιτροπής χαιρόμαστε για αυτή τη θετική ατμόσφαιρα εργασίας που διέπει το έργο του εισηγητή με τους σκιώδεις και αναμένουμε τις τροπολογίες συμβιβασμού σε σχέση με αυτά που άκουσα σήμερα, μιλάμε για ελάχιστη εναρμόνιση. Αυτή είναι και η παράγραφος 2 του άρθρου 1, η ουσία δηλαδή για την πρότασή μας για να κρατήσουν τα κράτη-μέλη το σύστημα που έχουν με άλλα πιο ευέλικτα κριτήρια. Αυτό θα πρέπει να το διασαφηνίσουμε κατά την έγκριση αυτού του κειμένου. Επίσης υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός σε όλα τα κράτη-μέλη, όπως ορίζει η οδηγία, η οποία μεταφέρεται στα κράτη-μέλη με ε, ε, ρήτρες διασφάλισης. Ε, σε σχέση με τους ειδικού όρους, ακούσαμε ότι θέλουμε να ενισχύσουμε συγκεκριμένα κριτήρια. Περιμένουμε προτάσεις, αλλά γνωρίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο τρόπος χρηματοδότησης αυτών των φορέων για να διασφαλίσουμε την διαφάνεια. Η Επιτροπή δεν θέλει να απαγορεύσει τις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις, διότι αποτελούν εχέγγυο της λειτουργίας του συστήματος, γιατί πολλές φορές αυτοί οι φορείς δεν διαθέτουν προϋπολογισμό. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνει υπό συνθήκες διαφάνειας, αποφεύγοντας ε, τη σύγκρουση συμφερόντων. Επίσης, άκουσα τι είπε ο εισηγητής σε σχέση με τις εξαιρέσεις τύπου Ombudsman. Θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό δηλαδή την ε, απομάκρυνση από οποιαδήποτε ε, ειδική ε, δικαιοδοσία. Ως προς το opt-in ή out, ξέρετε τη θέση μας. Θέλαμε να τηρήσουμε την αυτονομία των κρατών μελών ανάλογα με το τι επιλέγουν. Υπάρχουν υπέρ και κατά και στα δύο. Άρα θα πρέπει να κρατήσουμε την αυτονομία των κρατών μελών σε αυτό το τομέα και σε άλλους. Γιατί μιλάμε και για το δικαίωμα διαδικασίας, το οποίο επίσης θα πρέπει να τηρηθεί. Ως προς την ε, άγρα δοσιδικία στο forum shopping, ε, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι δική μας πρόταση η οποία θα οδηγήσει σε ένα άγριο φόρουμ shopping, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο δεν έχει αλλάξει. Πού θα γίνει λοιπόν η προσφύγη στη χώρα του εμπόρου ή στη χώρα όπου επέρχεται η ζημία ή η βλάβη. Η πρότασή μας δεν θα αλλάξει ως προς την επιλογή του ευνοϊκότερου δικαστηρίου. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για ε, την αναγνώριση αυτή και από τα άλλα κράτη-μέλη και έτσι μπορεί να γίνει προσφύγη εκπροσωπώντας ε, καταναλωτές πολλών ε, κρατών μελών. Είτε στο χώρο που κατοικεί ο έμπορος, κάτι το οποίο θα ήταν καλύτερο ίσως. Τώρα η αρχή ότι αυτός που χάνει πληρώνει, σε μία αιτιολογική σκέψη μιλάμε για αυτή την αρχή η οποία ισχύει σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο γιατί υπάρχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες στις οποίες αναφέρθηκε η κυρία Χαουτάλα αλλά καταρχήν θα πρέπει να έχει ισχύ. Αλλά διατηρώντας φυσικά την αυτονομία των κρατών μελών σε αυτό το τομέα. Ε, τώρα, σε σχέση με τα έξοδα έκτακτων αναγκών, contingency fees δεν προβλέπονται ε, δεν μιλάμε για μία οδηγία σε σχέση με τη σύσταση που υπήρχε σε σχέση με τις συλλογικές προσφυγές. Μιλάμε λοιπόν για αυτό το θέμα στην αιτιολογική σκέψη. Υπάρχει μία επιλογή που προβλέπεται εδώ για τα κράτη-μέλη. Αλλά το σκεπτικό που μας διέπει είναι να μην ενθαρρύνουμε αυτά τα έκτακτα έξοδα, γιατί δεν θέλουμε να γίνει εμπόριο ε, η διαφορά, να γίνει αντικείμενο εμπορίου η διαφορά. Θα πρέπει καταναλωτές να έχουν ένα άλλο μέσο το οποίο δεν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις συλλογικές προσφυγές για να υπάρχει καλύτερη διασφάλιση δικαιωμάτων χωρίς όμως καταχρήσεις. Είμαι στη, θέση του ε, στη διάθεση συγγνώμη, του εισηγητή και των σκιωδών και περιμένουμε αυτές τις τροπολογίες συμβιβασμού. Ευχαριστώ και σας. Πρέπει να πούμε ότι η έγκριση από την Επιτροπή έχει προβληθεί για τις 6 Δεκεμβρίου τώρα που βρίσκεται στην αίθουσα ο κύριος Φως, μπορούμε να επιστρέψουμε στο σημείο 29 της ημερήσιας διάταξης που αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την αναφορά με βάση αυτή την οδηγία. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο συγγνώμη που δεν ήμουν από αυτή τη στιγμή. Απλά χρειάστηκε να συζητήσω κάτι διαφορετικό. Έχουμε λοιπόν ήδη ολοκληρώσει δύο τριμερείς διαλόγους και μας απομένουν ακόμα τρεις τριμερείς διαλόγοι. Στις 26 του μήνα, μετά την επόμενη εβδομάδα 3 Δεκεμβρίου και μετά 13 Δεκεμβρίου τρίτη φορά. Ε, και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε και μία ακόμα μερομηνία για συνάντηση γιατί ουσιαστικά τέσσερις εβδομάδες μας απομένουν ακόμα και τα μεγάλα προβλήματα δεν έχουν ακόμα επιληθεί. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 11 και το άρθρο 13 θα κάνουμε μια περαιτέρω εις βάθος συζήτηση κατά την επόμενη συνάντηση του τριμερούς διαλόγου και παρόλα αυτά ε, ε, δείχνει δύσκολη να είναι μια προσέγγιση ανάμεσα στις διαφορετικές πλευρές. Τι έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα. Έχουμε καταφέρει για τα άρθρα 7 έως 10 κάποια πρόοδο σε ό,τι αφορά ε, για παράδειγμα τα out of commerce works αλλά και το video on demand και από εκεί και μετά έχουμε και τα άρθρα 14 έως 16α της έκδοσης του κειμένου από την πλευρά του Συμβουλίου, τα οποία θα συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα και έχουμε θέσει στους εαυτούς μας συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους θέλουμε να επιτύχουμε ακριβώς μέσα σε αυτές ε, σε αυτούς τους επόμενους τριμερείς ε, διαλόγους, έτσι ώστε τελικά να έχουμε και απτά αποτελέσματα και από εκεί και μετά να μπορέσουμε στο τέλος να εστιάσουμε πραγματικά στα ιδιαίτερα δύσκολα ζητήματα. Όλα αυτά βέβαια δεν θα είναι εύκολα και θα χρειαστεί να καταδείξουν σε οι πλευρές ε, με ορισμένη ευελιξία μια διαλλακτικότητα σε ό,τι αφορά τις λύσεις που θα βρούμε χωρίς ε, βέβαια αυτό να σημαίνει ότι τώρα πρέπει να αρχίσει κανείς να ανησυχεί ε, επειδή αναφερόμαστε ή αναφέρουμε τον όρο ευελιξία. Όχι, απλώς θέλουμε να φτάσουμε σε λύσεις οι οποίες θα ευθυγραμμίζονται με τα όσα έχουμε συμφωνήσει στο κείμενο του Κοινοβουλίου αλλά για να το επιτύχουμε θα πρέπει να είμαστε και λίγο πιο ανοιχτοί απέναντι στις προτάσεις που θα έρθουν από την άλλη πλευρά, χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε ακριβώς τι ακριβώς θα είναι αυτό, τι θα προκύψει. Και βέβαια να πω ότι οι τριμερείς διαλογές όπως οργανώνονται είναι πολύ σύντομοι για να επιτύχουμε αυτό που επιθυμούμε, αλλά αυτό που θα κάνουμε εμείς είναι θα προσπαθήσουμε σε σχέση με τους στόχους που θέσαμε να επιτύχουμε ό,τι μπορούμε και πραγματικά ας πούμε την επόμενη εβδομάδα θα παραμείνουμε στη συζήτηση έως ότου επιτύχουμε τον λόγο ε, στόχο. Και όπως είπα, μέχρι στιγμής ασχοληθήκαμε με τα άρθρα 7 έως 10 και θα ασχοληθούμε περαιτέρω με τα άρθρα 14 έως 16α της ε, εκδοχής του κειμένου του Συμβουλίου και από εκεί και μετά θα εστιάσουμε στα βασικά ζητήματα. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε εδώ να εστιάσουμε τελικά να περιορίσουμε ε, τη συζήτηση σε εκείνα που πραγματικά είναι πολύ σημαντικά. Εντάξει, μίλησα πολύ, δεν είπα πολλά πράγματα βέβαια, το γνωρίζω, αλλά σας λέω ότι δεν υπάρχουν απτά αποτελέσματα αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα υπαρκτά και πραγματικά σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή τη διάσταση απόψεων. Θα χρειαστεί περαιτέρω συζήτηση για να τα υπερκεράσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το κείμενο είναι δύσκολο, το γνωρίζουμε και όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και ο εισηγητής και οι σκιώδεις. Καταρχήν δυσκολίες από, τα, ε, από το ίδιο το κοινοβούλιο που δυσκολεύεται να μας βρει διερμηνής ή χρόνο στο σχεδιασμό ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι διερμηνείς. Αυτό το θεωρώ εντελώς απαράδεκτο. Εντελώς απαράδεκτο, διότι πρόκειται για ένα τρόπο να μας ε, εμποδίζουν για, επί ενός κειμένου πολύ δύσκολου, το γνωρίζουμε όλοι και οι σκιώδεις ακόμα περισσότερο και θα ήθελα κύριε Σιγητά αν ή δυνατόν σήμερα ή αν, αν μπορείτε αύριο εσείς πρέπει πάντως να το κάνετε, να στείλετε μια επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και να του πείτε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνουν συναντήσεις σκιώδων ή ακόμα περισσότερο τριμερείς διάλογοι χωρίς διερμηνία. Παραδείγματο χάρη, όταν ο φίλο μας, τον οποίο ε, σέβομαι, ο κύριο Έλμαρ Μπρόκ, ε, ζητά μία συνεδρίαση, βρέθηκαν για κάποιους που είναι σεβαστοί στο, στο κοινοβούλιο η απαραίτητη διερμήνηση. Αυτό δεν είναι ασήμαντο. Δεν μπορούμε να ε, στηριζόμαστε σε περίπου κατανόηση, γιατί εδώ διακυβεύονται χρήματα και θέματα. Υπάρχουν θέματα που ε, έχουν στραφεί εναντίον μας, εμάς, των μελών, μεγάλοι καπιταλιστές από την Καλιφόρνια, οι οποίοι ξεκινούν εκστρατείες ψεύδους, που δεν το κάνουν ούτε χειρότεροι βασανιστές, ας πούμε στις 5 Ιουλίου όταν χρειάστηκε να ψηφίσουμε για πρώτη φορά στην Ολομέλεια το κείμενο που εγκρίθηκε από την Νομική Επιτροπή που δεν το κάναμε χωρίς λόγο μας είπαν ότι δεν μας αφορά το κείμενο και γράφει το κείμενο ότι επιτρέπεται μία εκστρατεία επιτράπει μία εκστρατεία για να ζητούν να καταψηφιστούν τα πνευματικά δικαιώματα. Επειδή ήταν όργανο λογοκρισίας, θα τη Wikipedia και όταν ψάξαμε λίγο περισσότερο να δούμε τι κρύβεται, διαπιστώσαμε ότι ήταν το Ίδρυμα Google που είχε πληρώσει την όλη αυτή υπόθεση. Μας συμπεριφέρονται άσχημα γιατί οι ίδιοι λομπι, λομπίστες παρεμβαίνουν στους υπολογιστές μας χιλιάδες μηνύματα εντός λίγων ωρών και πιστεύω ότι πρέπει το Κοινοβούλιο να διαμαρτυρηθεί για να υπερασπιστεί τα μέλη του, για να μπορούμε να λειτουργούμε ελεύθερα. Δεν είμαι φυσικά αγαθός, γνωρίζω το βάρος που έχει η καλλιτεχνική δημιουργία στην Ευρώπη με όλα αυτά Είμαστε πάνω από το, τα 540 δις το χρόνο. Το ακούσατε, 540 δις το χρόνο. Ότι εργάζονται εκατομμύρια άνθρωποι, περισσότερο δηλαδή από ότι στις τηλεπικοινωνίες και στην αυτοκινητοβιομηχανία και ότι αυτό βεβαίως πονάει τη Wall Street. για να μείνουν κάποια ε, δισεκατομμύρια στην ε, Ευρώπη και μας κακομεταχειρίζονται γιατί εδώ και δύο-τρεις μέρες το, η Google και οι θύνοντες άλλ, από άλλους οργανισμούς, άλλες πλατφόρμες επί, απειλούν ότι θα κόψουν την υπηρεσία ειδήσεων αν ε, περάσουμε περιορισμούς με την καουμπόικη, κλασική καουμπόικη νοοτροπία που προσπαθούν να επιβάλλουν όταν δεν μπορούν να κάνουν Αν ήταν εδώ ο κύριος Πασκουάλ θα θυμόταν και αυτός, γιατί ξέρω γιατί μιλάνω, μιλάω, ότι η, η Google κόντεψε να σκοτώσει την ΕΛΠΑΗ στην Ισπανία, αρνούμενη να, πληρώσει Επίσης, μας κακομεταχειρίζονται και αυτό είναι χειρότερο ε, για μένα γιατί γίνεται εδώ, γιατί αν δούμε το βάρος του lobbying, του βίαιου lobbying που ασκούν αυτές οι επιχειρήσεις, θα ήθελα να μας πει ο εισηγητής, και δεν κάνω δίκη σκοπό ε, ε, προθέσεων, γιατί μετά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, η οποία έγινε με, επί τη βάση του κειμένου που εμείς εγκρίναμε και που είχαμε εντολή και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, είναι κυρίαρχη η Ολομέλεια, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το οποίο ψήφισε, γιατί συνεχίζουμε να, να λαμβάνουμε, όπως και εσείς κύριε Σιγητά, αυτούς τους λομπίστες, το YouTube συγκεκριμένα, την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο, στο τραπέζι σας, μετά από πρόσκληση δική σας, είχατε και βουλευτές, απολύτως δικαιωμά σας φυσικά, πολλοί αρνήθηκαν να πάνε ήμουν και εγώ, δεν θα, βάλω, δεν θα πατήσω εκεί που υπάρχουν αυτοί. Όταν βλέπουμε ότι στις συζητήσεις μας έχουμε τους, τους τρί, τα τρία θεσμικά όργανα, όχι τους ξένους, τους τρίτους καπιταλιστές, βλέπω ότι η ψηφοφορία είναι κυρίαρχη. Δεν μπορούμε να συζητάμε με τα λόμπι αφού μας έδωσε την εντολή του το Κοινοβούλιο, η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Και επιπλέον οι συνάδελφοι, οι βουλευτές που πήγαν, ένας παρευρίσκεται, εντυπωσιάστηκαν, θέσουν, θέτουν ερωτήσεις στον Chief Executive Officer της συγκεκριμένη εταιρεία από την Καλιφόρνια και δεν έλαβαν απάντηση. Τους ε, συμπεριφέρθηκαν σαν να ήταν ανύπαρκτοι. Προσπαθώ να καταλάβω λοιπόν, κύριε Σιγητά, τι επιδιώκεται προσκαλώντας αυτούς τους ανθρώπους σε μια διαθεσμική περίοδο που δεν θα έπρεπε κατά τη γνώμη να βρίσκονται. Και επίση, επειδή είμαι εδώ σχεδόν 15 χρόνια, αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ, είναι άνευ προηγουμένου. Αν πρόκειται να θεσμοθετηθεί, ε, πρέπει να πω ότι είσαστε ο, ο, ο Επίσης, πρέπει να ζητήσω από τους συναδέλφου να να αντιμετωπίσουν τα θέματα με ισότητα. Η κυρία Χανιμπόλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ακούστηκε, το θέμα ήταν εξαιρετικά δύσκολο εξ αρχής. Εντελώς πολλωμένες απόψεις. Στα 20 χρόνια ποτέ δεν έχω ξαναδεί τέτοια έκθεση. Οπότε τώρα θεωρώ ότι ο εισηγητής και εμείς οι ευρωβουλευτές έχουμε την τεράστια ευθύνη να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο, ότι αυτό το οποίο πέρασε θα το υπερασπιστούμε και ότι θα λειτουργήσει. Η δεύτερη, με τη δεύτερη προσπάθεια ε, πέρασε με πάνω από 200. Ήταν μεγάλη πλειοψηφία. Φυσικά, μόλις μεταβίας πέρασε από την Επιτροπή μας. Όμως τελικά ήταν ουσιαστική, ήταν σημαντική η πλειοψηφία η οποία κατέληξε μετά από διαπραγματεύσεις. Πρέπει, μπορούμε να πούμε ότι σε, με μεγάλη πλειοψηφία το Κοινοβούλιο το υποστήριξε και είναι σημαντικό να το κάνουμε αυτό. Ο κύριος Καβαντάς μίλησε για τους λομπίστες. Εγώ δεν ήμουν εκεί φυσικά, αλλά άκουσα, ε, έφτασαν στα αυτιά μου ε, η παρουσία των λομπιστών και τι προσπαθούν να κάνουν αυτοί στο Κοινοβούλιο. Προσπαθούν να ξοδέψουν χρήματα και χρόνο και πολλά επιχειρήματα που σε πολλές περιπτώσεις δεν ευσταθούν για να πείσουν τον κόσμο να κάνει αυτό που επιθυμεί η Google και οι άλλες πλατφόρμες. Πρέπει να, το αντιμετωπίσουμε αυτό, γιατί εσείς είστε καθοριστικός στο να περάσει αυτό από το Κοινοβούλιο και βεβαίως είναι δουλειά σας να συνεχίσει. Είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό να ε, να σταθούμε για να φροντίσουμε ότι θα ε, ισχύσει αυτό που ψήφισε το Κοινοβούλιο. Θα υπάρχει πίεση για αλλαγή και ξέρετε κάποιες ελάχιστες αλλαγές αλλάζουν πολλά πράγματα. Για μένα κάτι που προτάθηκε αφορά το value gap, το κενό αξίας, το χάσμα αξίας η πλατφόρμα θα πρέπει να έχει ευθύνη. Λένε μερικές φορές ή να είναι λίγο, να έχει λίγη ε, αστική ευθύνη κλπ. Όχι για πάντα. Είναι όλα αυτά υπονόμευση. Είναι πολύ σημαντικό για τα σημαντικά, για αυτά που είναι ουσιαστικά εδώ, να επιμείνουμε στη γραμμή του Κοινοβουλίου, που ε, ήταν δύσκολο, με δυσκολίες επιτεύχθη. Ξέρω ότι θα υπάρχουν έχουν δυσκολίες γιατί η Google και οι άλλοι θα φτάσουν στο Συμβούλιο. Έχουν ε, ε, χρήματα για να συνεχίσουν την εκστρατεία τους. Δεν πρόκειται να είναι εύκολα τα πράγματα και θα γίνουν ακόμα δυσκολότερα αν δεν υπάρξει σωστή μετάφραση και αν οι συνεδριάσεις δεν, ε, έχουν αρκετό χρόνο και αρκετά, δεν είναι αρκετά σαφείς. Βλέπω εδώ μια συνωμοσία για να δυσκολεύσουν οι διαπραγματεύσεις τα, τα μέλη της Επιτροπής θέλουν να σας υποστηρίξουν, όπως και οι σκιώδεις, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αφήσουμε να υπονομευθεί αυτή η προσπάθεια. Είναι κάτι που επιθυμούν στο Κοινοβούλιο και η ευθύνη μας είναι να φροντίσουμε να περάσει από τους τριμερείς διαλόγους, όπως το ψήφισε το Κοινοβούλιο. Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε, δεν θα η θέση μου παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα. Γιατί εγώ είμαι από αυτούς που έχασαν στα πλαίσια της εντολής στην ψηφοφορία για λόγους που ο Ζαμαρί Καβαντά γνωρίζει πολύ καλά. Υπάρχει διαφορά ουσίας ε, μεταξύ μας. Και επιμένω να λέω ότι η, η εντολή ε, δεν είναι όπως θα την ήθελα. Όμως θα ήθελα να υποστηρίξω τον Ζαν Μαρί Καβαντά επί της ουσίας. Βρισκόμαστε στα πλαίσια της θητείας μας και στα πλαίσια της θητείας και εντολής θα πρέπει να, λύσουμε, να τηρήσουμε την δημοκρατική εντολή. Ε, αν ήμουν εισηγητής θα υποστήριζα το Κοινοβούλιο. Είδα ότι έγινε άλλες φορές στην ΙΜΚΟ από τον πρόεδρο της Επιτροπής που αν και μειοψηφούσε υποστήριξε το κείμενο για το οποίο είχε εντολή. Δεν είναι αυτή η θέση μου, όμως το Κοινοβούλιο θα πρέπει να υποστηριχθεί διότι έχει μία θέση την οποία θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Ε, έναντι των λόμπιστ, όποιοι και να είναι αυτοί, δεν θα πρέπει να τους συναντάμε τη στιγμή που έχει θεσμοθετηθεί η θέση μας ή να δεχτούμε όλους τους λόμπις πριν λάβουμε απόφαση. Γι' αυτό υποστηρίζω τον Ζαμαρί Καβαντά ως προς το θέμα της δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Um, <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω ευχαριστώντα τον συνάδελφο Αξελπού για ε, την... το ε, τεράστιο έργο που έχει αναλάβει για λογαριασμό όλων μας ε, εδώ, σε αυτή την Επιτροπή, ανεξαρτήτως του ποια θέση πρεσβεύουμε στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση. Και δεν νομίζω πως θα μπορούσαμε να συμφωνούμε όλοι μας σε σχέση με όλα τα ζητήματα. Υπάρχουν δηλαδή διαφορετικά επιχειρήματα που ε, υποστηρίζουν διαφορετική από εμά και διαφορετικές συμμαχίες έχουν σημαντιστεί για διαφορετικά ζητήματα. Πάντως, θα πρέπει πραγματικά να αναγνωρίζουμε ε, τη δουλειά που κάνει και έχει κάνει ο κύριος Σεβός για λογαριασμό της δικής μας Επιτροπής και θα πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου. Δεύτερο που θα ήθελα να αναφέρω. Εγώ παρευρέθην στο συγκεκριμένο γεύμα και ο λόγος για τον οποίο παρευρέθην ήταν ότι Γνωρίζω βέβαια ποια είναι η ιδέουσα διαδικασία και τι ήθιστε να συμβαίνει και εδώ και αλλού. Ε, πάντως, επαναλαμβάνω, ε, το παρευρέθην γιατί θεώρησα πως ήταν μια ευκαιρία να βρεθώ στην ίδια αίθουσα και να ακούσω από την άλλη πλευρά του τραπεζιού μία από τις πλατφόρμες η οποία είχε συμμετάσχει και είχε πάρα πολλές σχέσεις με αυτό εδώ το κοινοβούλιο ε, με διαφορετικούς τρόπους. Και η πλατφόρμα αυτή ήταν παρούσα ε, και δραστηριοποιούνταν κατά όλη τη διάρκεια της συζήτησης που γινόταν εδώ σε αυτό το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και η επίδραση, αν θέλετε, που είχε εδώ δεν γινόταν άμεσα με το δικό μας κοινοβούλιο, αλλά μέσω ακριβώς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως ε, το έχουμε δει δηλαδή εδώ και πραγματικά υπήρξε ένας βομβαρδισμός, πραγματικός βομβαρδισμός με διάφορες δράσεις τύπου lobbying η πλειοψηφία των οποίων αυτών δράσεων και μηνυμάτων ήταν, ε, περιείχε λανθασμένες πληροφορίες. Εγνωρίζουμε πώς ε, λειτουργούν τα πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιος λαμβάνει μία είδηση, ε, δίνει τη δική του ερμηνεία σε αυτή την είδηση και την μεταβιβάζει στον επόμενο, ο οποίος την ερμηνεύει και αυτός με τη δική του πλευρά και ούτω καθε Και τελικά καταλήγουμε σε κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες απηχούνται με τελείω διαφορετικό τρόπο, ε, άσχετο με τον τρόπο με τον οποίο εμεί πρεσβεύουμε τα πράγματα, ποια είναι η δική μα θέση. Άρα λοιπόν, για πρώτη φορά ε, είχα τη δυνατότητα να θέσω συγκεκριμένα ερωτήματα σε μία από αυτές τις συγκεκριμένες πλατφόρμες ε, και δεν ε, είδα καμία, μα καμία πραγματικά διάθεση πραγματικής ε, συναλλαγής από την δική τους ε, πλευρά. Αν λοιπόν κάποια από αυτές τις πλατφόρμες θεωρούσε ότι ερχόμενοι σε επαφή μαζί μας με αυτόν τον τρόπο προκειμένου να επηρεάσουν κατά κάποιο τρόπο την πώς θα εξελιχθεί η συζήτησή μας, το μόνο που κατέδειξε είναι την τρομερή αφέλειά τους. Έχουμε προχωρήσει αρκετά σε σχέση με τη διαδικασία διαλόγου, σε σχέση με αυτή την πρόταση. και δεν νομίζω πως υπονομεύεται με κάποιο τρόπο η αξιοπιστία της διαδικασίας ε, η οποία έχει ξεκινήσει και τρέχει μέχρι στιγμής. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει δηλαδή να γίνει εκτεταμένη συζήτηση που συζητήσεις ενδεχομένως μπορούν να έχουν λάβει ή όχι χώρα. Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι και ε, ε, δεσμευόμαστε οι ίδιοι σε ό,τι αφορά την δέουσα διαδικασία που προβλέπεται στο Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο και έχει προβληθεί και τα θεσμικά μας όργανα. Thank you very much, Mr. Chair. I think... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το οποίο καθίσταται όλο και πιο εμφανές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε για να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς και τα πιο αμφιλεγόμενα άρθρα του κανονισμού είναι ότι πρέπει να ακούσουμε περισσότερο την πανεπιστημιακή εμπειρογνω... τους πανεπιστημιακούς εμπειρογνώμονες που έχει προσφερθεί στο Κοινοβούλιο από πάρα πολλά ανεξάρτητα πανεπιστήμια που έχουν ε, δραστηριοποιηθεί Επίσης, τα Ινστιτούτα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που έχουν σχολιάσει και που έχουν ε, προσφέρει τα θέματα της δευτερογενούς αστικής ευθύνης και άλλα. Ε, πολλές δηλαδή ε, πολλές επικοδομητικές συμβαστικές προτάσεις από τον πανεπιστημιακό χώρο. Επίσης, αυτό καθίσατε σταφές εκ του ότι η Google παλεύει για να γίνουν υποχρεωτικά τα upload filters. Δηλαδή αυτοί ε, οι πολίτες που γράφουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο κατά του, ε, των upload filters έχουν ε, λάθος τη θεωρηθεί ότι το έκαναν με δόλο, διότι μια εταιρεία που χρησιμοποιεί το upload filter δεν θα έχει αστική ευθύνη. Αυτό θα το έκανε ε, άχρηστο. Δηλαδή θα ε, διέδιδε ακόμα περισσότερο τη χρήση αυτών των φίλτρων και δεν θα ε, άφηνε, δεν θα διεύρυνε την προσφορά. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε μια απόσταση, να δώσουμε χρόνο, να μελετήσουμε τις προτάσεις των πανεπιστημιακών για να προχωρήσουμε. Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να αποφθηνόμαστε σε μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και μέσων ενημέρωσης για να συμβιβαστούν μεταξύ τους, γιατί ένα τέτοιο συμβιβασμός δεν θα λάβει υπόψη του το δημόσιο συμφέρον και τους ψηφοφόρους μας που μας ζητούν να υπερασπιστούμε τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Uh, Ωραία. Κύριε Φως, θέλετε να πάρετε το λόγο και πάλι παρακαλώ. Γνωρίζουμε όλοι μας ότι η διαδικασία αυτή είναι πάρα πολύ περίπλοκη. Ε, είναι λίγο ταμένα τα αισθήματα. Η συζήτηση τη μία στιγμή κινείται προς τη μία κατεύθυνση, την άλλη στιγμή κινείται προς την άλλη κατεύθυνση, οπότε θα πρέπει όλοι να ερεμήσουμε λίγο και να δούμε τι ακριβώς θέλουμε να επιτύχουμε. Νομίζω πως είναι σαφέστατο το τι πρέπει να επιτύχουμε. Έχουμε μία εντολή που έχουμε λάβει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχει από την απέναντι πλευρά το Συμβούλιο με τη δική του εντολή. Και τώρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο κάπως να βρούμε έναν τρόπο να συμβιβάσουμε αυτές τις δύο εντολές μεταξύ τους. Ε, ε, επιχαίρω το γεγονός ότι η εντολή αυτή δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία και γι' αυτό σε σχέση με τα άρθρα 11 και 13 ακολουθώ και την αντίστοιχη γραμμή. Ωστόσο, είτε αυτή η εντολή ισχυρή είτε όχι, να συνδιαλλαγούμε με τους άλλους θα πρέπει να συμβεί. Είτε αυτοί οι άλλοι συνδιαλασσόμενοι είναι οι πλατφόρμες, είτε οι χρήστες, είτε ε, απέναντι πλευρά, το Συμβούλιο. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακούσουμε τις δικές τους αντιδράσεις, τις δικές τους απόψεις ως προς το τι ακριβώς θεωρούν σε σχέση με το με την κάθε λύση, έτσι ώστε να φτάσουμε στην κατάλληλη λύση. Δεν μπορούμε δηλαδή να βρούμε λύση εάν σε όλα τα επίπεδα είμαστε ακριβώς, ε, απλώς και μόνο αντιπαραθετικοί. Ε, ε, δηλαδή δεν μπορούμε απλώς και μόνο να πρεσβεύουμε τη δική μας άποψη αποκλείοντας κάθε δυνατότητα εξέβρεσης ενός συμβασμού με την άλλη πλευρά. Εάν κάποιος δεν θέλει να έρθει σε επαφή με κάποιον άλλον, μπορεί να το κάνει. Ωστόσο, θεωρώ πως με περισσότερο επικοινωνία μπορούμε να επιτύχουμε και περισσότερη κατανόηση, αν θέλετε, της όλης διαδικασίας. Γιατί είμαστε, νομίζω, πως ο τέταρτος player, ο τέταρτος παίκτη σε αυτήν την συνδιαλλαγή ή σε αυτήν την επικοινωνία, σε αυτό το διάλογο, ο οποίος πραγματικά είναι ο πιο διαλλακτικός, που έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με όλους. Ε, και νομίζω πως αυτά που έλαβαν χώρα στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα ήταν θετικά γιατί ακούσαμε τελικά τα προβλήματα που αυτή η άλλη πλευρά δηλαδή αντιμετωπίζει οι πλατφόρμες και ούτω καθεξής. Ε, τώρα το κατά πόσο συμφωνούμε ή όχι είναι άλλο θέμα αλλά καλό είναι να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. και είναι χρήσιμο για παράδειγμα αυτό που κάναμε να ακούσουμε τα προβλήματα από την πλευρά των χρηστών όπως έγινε δηλαδή πριν από το ε, καλοκαιρινό διάλειμμα. Είναι καλό λοιπόν να γνωρίζουμε όλα τα προβλήματα έτσι ώστε να δούμε ποια θα είναι τελικά η καταλληλότερη λύση. Όμω, δεν θα πρέπει να είμαστε έτσι συναισθηματικά φορτισμένοι, αν θέλετε, ε, και να λέμε στο πλαίσιο αυτή τη διαδικασία, Όχι, αυτό δεν το δέχομαι, το άλλο δεν το δέχομαι. Θα πρέπει αντιθέτω να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση η οποία από τη μία πλευρά δεν καταπνίγει, αν θέλετε, την ψηφιακή εξέλιξη, αλλά και από την άλλη πλευρά εμ, θέτει τους κατάλληλους περιορισμούς και προστατεύει με τον κατάλληλο τρόπο τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή αυτό είναι το καθήκον μας, ε, να επιτύχουμε λοιπόν μια ισορροπημένη λύση ακριβώς ε, βρίσκοντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στα διαφορετικά συμφέροντα. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ε, αυτό το καθήκον μου, αντιλαμβάνομαι την ευθύνη που αναλαμβάνω, ειδικότερο σε ό,τι αφορά τα άρθρα που συζητούνται αυτή τη, σε αυτή τη φάση και θα πρέπει να δούμε πώς θα πάνε τώρα τα πράγματα στο πλαίσιο της συζήτησης με το Συμβούλιο. εντάξει, στο τέλος μπορεί το όλο εγχείρημα να αναβαγίσει. Αλλά προς το παρόν ας μην ε, αγκιστρωνόμαστε σε συγκεκριμένα ε, ζητήματα ε, λέγοντας ότι δεν επαναχωρούμε σε τίποτα. Ας δούμε ποια θα μπορούσε να είναι μια εφικτή λύση και θα ήθελα να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε αυτή τη λύση ως τις 13 και στις 14 Δεκεμβρίου. Γιατί τα πράγματα δεν πρόκειται να βελτιωθούν από μόνα τους. Έχουμε κάνει διαξωδικέ συζητήσει εδώ και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ διαφορετικών στοιχειωδών εισηγητών και έχουμε ακούσει διαφορετικέ λύσει. Από τη μία εκείνες δηλαδή που είναι, κινούνται περισσότερο προ την ψηφιακή πλευρά, άλλε οι οποίε δίνουν περισσότερη έμφαση στα δικαιώματα ε, πνευματικής Οπότε ε, θα πρέπει να δούμε πού μπορούμε να βρούμε μια λύση όσο και αν αυτή είναι δύσκολη. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μα ότι κανεί δεν θα επιτύχει στο 100%, ε, 100 στο ακέραιο δηλαδή την ικανοποίηση των αξιώσεων του, ούτε εκείνοι οι οποίοι είναι οι διοκτήτες των ε, δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία, ούτε οι χρήστε χρήστες ούτε κανείς. Ε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ανοιχτή στάση, μια διαλλακτική στάση, να δούμε ποια είναι τα όρια και πώ μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Γιατί αν δεν λειτουργήσει μια τέτοια μέθοδο διαλόγου, δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Δηλαδή, αν αναμείνουμε τρία-τέσσερα χρόνια ακόμα, τα πράγματα θα έχουν εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, θα έχουν μεταβληθεί, αν θέλετε, οι συσχετισμοί δυνάμεων και έτσι τα πράγματα θα είναι πιο περίπλοκα. Ε, κάτι που ανέφερε σωστά ο συνάδελφος Καβένα είναι το ότι μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να είμαστε και ευέλικτοι σε ό,τι αφορά τις διαφορετικές συναντήσεις που προβλέπονται, είτε σε επίπεδο ε, σχεδόν εισηγητών, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ανταποκρίνεται στη δομή που προβλέπουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό δηλαδή της ε, διαρμηνίας. Σε κάποιες δηλαδή περιπτώσεις η υπηρεσία διαρμηνίας δεν μας δίνει τη δυνατότητα ε, να έχουμε κάποια συνεδριάσει με ερμηνεία. Στη συγκεκριμένη τώρα περίπτωση, σε αυτή τη συζήτηση, βρισκόμαστε υποχρονική πίεση. Και δεν είναι πίεση έξωθεν, είναι όρια χρονικά τα οποία έχουμε θέσει εμεί στου εαυτού μα ε, Και ακριβώ είπα ότι ε, στο πλαίσιο αυτής της ευελιξίας, ακριβώς επειδή θέλουμε να βρούμε μια λύση, θέλουμε περισσότερο τριμερή διάλογο, προκύπτει αυτό το πρόβλημα το ότι δηλαδή δεν έχουμε την διαρμηνία πάντοτε εκεί που το θέλουμε, ακριβώ γιατί δεν βασιζόμαστε στη συνείδη ε, οργάνωση των εργασιών με τη διερμηνία. Και εμένα θα μου άρεσε περισσότερο όλε οι συναντήσει αυτέ να καλύπτονται και με διερμηνία, γιατί όπω είπε και σωστά ο κ. Κάπατρα, υπάρχουν ορισμένε φορέ συγκεκριμένε χρειέ του κειμένου, ε, οι οποίε δεν γίνονται κατανοητέ, δεν περνούν με τον ίδιο τρόπο σε άλλη γλώσσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω ότι παρόλα αυτά βρισκόμαστε σε μια άγουσα που μπορεί να μας οδηγήσει σε κοινέ λύσει. Δηλαδή, αν λειτουργεί ένα κείμενο σωστά, τότε θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να λέμε καλό σας ξανασυναντηθούμε για να το ξανασυζητήσουμε και να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπροστά. Έτσι προσεγγίζω τουλάχιστον εγώ αυτήν την όλη αυτή τη συζήτηση. Ούτω ή άλλω το να καταλήξουμε σε αυτή τη θέση από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα και νομίζω πως θα πρέπει ε, πράγματι να συζητήσουμε κάποια στιγμή αυτήν την ισχύ που αρχίσουν να αποκτούν τέτοιου είδου πλατφόρμες, πλατφόρμες δηλαδή οι οποίες ανά πόσο στιγμή μπορούν να δημιουργήσουν ε, ε, μια κρίσιμη μάζα αν θέλετε η οποία κάνει μια προσπάθεια να επηρεάσει οποιαδήποτε ε, νομοθετική διαδικασία, οποιαδήποτε συζήτηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αρχίσουμε να κινούμαστε προς μια απτή ε, λύσεις. Δεν οδηγεί εδώ δηλαδή πουθενά το να ε, πανικοβαλόμαστε ή το να αγκιστρωνόμαστε σε συγκεκριμένες θέσεις. Θα πρέπει να δούμε πώς συστηματικά μπορούμε να προσεγγίσουμε μια λύση. Ευχαριστώ. Point number Λοιπόν, ευχαριστώ. Μπορούμε πιστεύω να κλείσουμε το 29 όσον αφορά το 31. Έχουμε Έχουμε τα σημειώσεις του συγγητή του κυρίου Κοφεράτη, τα οποία ο κύριος Κοφεράτη ε, δεν μπόρεσε να, να παρευρεθεί και ζητά συγγνώμη. Θέλει να ευχαριστήσει τους συναδέλφους που υπέβαλαν 69 τροπολογίε στην έκθεσή του γιατί ε, διαπιστώνουμε ένα σημαντικό και επικοδομητικό στοιχείο που θα ενισχύσει και θα συμπληρώσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Όπως γνωρίζετε, το θέμα είναι σημαντικό στοιχείο της διακρατικής ε, δικαστικής διαδικασίας σε αστικά και εμπορικά ζητήματα και γι' αυτό στόχος της, της πρότασης της Κομισιόν είναι να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ταχύτητα της ε, επίδοσης των δικαστικών και εξοδίκων εγγράφων με και με ε, ηλεκτρονικές διαδικασίες. Στην έκθεση επιμένουμε στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων των εμπλεκομένων και οποιαδήποτε νέα ε, διαδικασία εισαχθεί να ε, εξασφαλίσει απρόσκοπτη και υψηλό επίπεδου ανταλλαγή εγγράφων και την ασφάλεια ε, συμφωνούμε με την πρόταση της εισαγωγής της ηλεκτρονικής επίδοσης των εγγράφων, όμως έχουμε προσθέσει ρήτρες ασφαλείας, κυρίως όσον αφορά το ότι ο αποδέκτης αποδέχεται αυτού του είδους την υπηρεσία. Για τα θέματα αυτά έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες προς την ίδια κατεύθυνση, οι οποίες ενισχύουν το κείμενο με θετικό τρόπο. Θεωρούμε ότι για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, το κόστος ε, των αυτών οι οποίοι ετούνται ε, την ε, ε, ε, ετούνται τις υπηρεσίες αυτές δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικό. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα ανώτατο όριο στην πληρωμή στο κόστος που μπορεί να επιβάλλουν τα κράτη-μέλη. Επιπλέον θεωρούμε ότι τα μέρη που έχουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος μέλους θα, μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν εκπρόσωπο ε, στο, ε, μέλο κράτος μέλους του δικαστηρίου. Η, επί των θεμάτων αυτών δεν είχαμε σχόλια και ελπίζουμε ότι η πρόταση μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω και να έχει ευρύ υποστήριξη από τους άλλους συναδέλφους. Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να καταλήξουμε σε, μια, ε, καλή, ε, σε ένα καλό αποτέλεσμα κατά την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Ράδιεφ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κοφεράτη για την έκθεση αυτή. Η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί βελτίωση και επίσπευση της υποβολής και λήψης των δικαστικών και εξοδίκων εγγράφων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις οι κανόνες επίδοσης των εγγράφων θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ταχεία και ασφαλή ε, παραλαβή τους και θα πρέπει να υπάρξει αποδεικτικό παραλαβής. Η πρόταση εισαγωγή της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των αρχών με τη δημιουργία ενός ε, αποκεντρωμένου συστήματος πληροφοριών η αποτελεί καλή και αξιόπιστη μέθοδο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη σύγχρονη τεχνολογία. Παρά τα αυτά, θα πρέπει να διευρυνθεί και να ενθαρρυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή. Θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη της ταχυδρομικής και επίδοσης και επίδοσης με ε, courier. Να εξασφαλιστεί ότι τα έγγραφα και, και τα, οι άλλες κοινοποίησεις είναι αληθή και ότι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της παραλαβής αποδεικνύει ότι ο παραλήπτης τα έχει λάβει και μάλιστα συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό ισχύει για έγγραφα που έχουν ληφθεί τόσο ε, σε φυσική μορφή, σε χαρτί, όσο και ηλεκτρονικά. Θα είναι σημαντικό, πιστεύω, ο παραλήπτης να μπορεί να αρνηθεί οι ε, έγγραφα που έχουν ε, υποβληθεί ηλεκτρονικά και έχω υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι το κόστος που θα προκύπτει όταν οι ειδικοί των δικαστηρίων οι άλλοι αρμόδιοι χρεώνουν κάτι το οποίο όμως δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικό και πρέπει να μελετηθεί με προσοχή ποιο θα είναι το ποσό. Πρόεδρος, δεν βλέπω να ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Μήπως θέλει η Κομισιόν να πάρει το λόγο. Όχι. Οπότε, στο σημείο αυτό, μπορούμε να πούμε ότι, ότι τελειώσαμε η έγκριση στην Επιτροπή θα γίνει στις 6 ή στις 10 Δεκεμβρίου. Δεν είμαστε ακόμα σίγουροι. Οπότε, συνεχίζουμε με το σημείο 32, μελέτη των τροπολογιών για τη συνεργασία μεταξύ δικαστηρίων των κρατών μελών για την διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις και έχει το λόγο ο κύριος Ράντζεφ ως συγητής. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι στιγμής δεν μπορέσαμε να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού, οπότε θέλω να επισημάνω κάποια από τα βασικά σημεία ο, ο χώρος της δικαιοσύνης απαιτεί δικαστική συνεργασία που ξεπερνά τα εθνικά σύνορα. Για το σκοπό αυτό και για να διευκολύνουμε την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει νομοθεσία για τη συνεργασία κατά την διεξαγωγή αποδείξεων. Το θέμα αυτό είναι κρίσιμη σημασία για την ρύθμιση της αμοιβαίας δικαστικής συνεργασίας σε ε, θέματα σε υποθέσεις αστικές ή εμπορικές μεταξύ κρατών μελών πρέπει ε, να αποτελεί το επαρκές ε, πλαίσιο συνεργασίας των κρατών μελών διακρατικά. Η η απόφαση του 2001 αποτελεί ε, το, το μέσο για να διεκπεραιώνονται ταχαίως οι τέτοιου είδους υποθέσεις και ξεκαθαρίζει και το ε, περιεχόμενο αυτών των ετοιμάτων. Επίσης θεσπίζει ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δικαστηρίων, πράγμα που επιτρέπει την άμεση ε, διεξαγωγή αποδείξεων στα δικαστήρια άλλων κρατών μελών. Πιστεύω ότι η πρόταση της Κομισιόν έρχεται σε κατάλληλο χρόνο και αποτελεί μια καλή ανταπόκριση στο πρόγραμμα REFIT. Είναι σημαντικό τα δικαστήρια των κρατών μελών να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία με σκοπό την επιτάχυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Κάτι τέτοιο δεν θα είναι δυνατόν αν δεν προσαρμοστούν οι κανόνες για τη διεξαγωγή αποδείξεων, κυρίως σε διαμεθοριακές περιπτώσεις. Η πρόταση της Κομισιόν θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω. Πιστεύω ότι και εγώ αλλά και άλλοι συνάδελφοι που έχουμε υποβάλει προτάσεις τροπολογιών ε, προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε κινηθεί. Όσον αφορά ας πούμε τον ορισμό του δικαστηρίου πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι πρέπει να αποδεχτούμε και άλλες οντότητες ε, πέρα των δικαστηρίων που είναι αρμόδιες στα διάφορα κράτη-μέλη για την ε, διεξαγωγή αποδείξεων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ε, τεχνολογική ουδετερότητα. Δηλαδή η, θα πρέπει να μην χρησιμοποιηθεί ο όρος video conference αλλά η τεχνολογία επικοινωνίας εξ Επίσης πρέπει να ε, διευκρινιστεί ότι η τεχνολογία επικοινωνίας εξ αποστάσεως ε, να εξασφαλίζει το επαγγελματικό απόρριτο και το προνόμιο του νομικού επαγγέλματος. Έχουν υποβληθεί τροπολογίες από αυτού. Όσον αφορά την πρόταση που επιτρέπει το ε, κάνει ε, διεξαγωγή αποδείξεων στο διπλωματικό προσωπικό θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη Σύμβαση της Βιέννης των Διπλωματικών Σχέσεων του 1961. Κατά την διεξαγωγή αποδείξεων, οι συμμετέχοντες σε μια video conference ή αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν άλλου είδους τεχνολογία θα πρέπει να έχουν επαρκή ενημέρωση για το χρόνο, τις συνθήκες αλλά και τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί κατά την υποβολή ε, αποδείξεων και υπάρχουν σχετικές, έχουν υποβληθεί σχετικές τροπολογίες. Η, επικοινωνία, η τεχνολογία της επικοινωνίας εξελίσσονται ταχύτατα και είναι σημαντικό να υπάρχουν τα προσωπικά στοιχεία. Η έκθεση καλύπτει κάποιες, με κάποιες τροπολογίες το θέμα. Η, η, ημερομηνία, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών έληξε στις 24 Οκτωβρίου λάβαμε 84 ε, σχετικές τροπολογίες και θα προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες να μπορέσουν να ψηφιστούν στην Επιτροπή στις 6 Δεκεμβρίου και στην Ολομέλεια στο τέλος Ιανουαρίου. Μήπως θέλει το λόγο, να πάρει το λόγο η Κομισιόν, από ό,τι βλέπω όχι. Χαιρετίζω την ομάδα των Τσέχων φοιτητών και τους καθηγητές τους που μας επισκέπτονται σήμερα. Στο σημείο αυτό μπορεί να, να λήξει το, η συζήτηση για το θέμα 32. Η, παρίσταται η κυρία Νίμπλερ, οπότε μπορούμε να επιστρέψουμε στο θέμα 28 και να ακούσουμε την παρουσίασή της του θέματος του πλαισίου προληπτικής αναδιάρθρωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά. Μέχρι στιγμή έχουν λάβει χώρα δύο τριμερεί διάλογοι σε ό,τι αφορά την προληπτική αναδιάρθρωση και τη δεύτερη ευκαιρία κατά τι επιχειρήσει. Αυτοί οι τριμερεί διάλογοι έτρεξαν ε, όπω αναμενόταν. Εμεί δηλαδή από την πλευρά του Κοινοβουλίου αναφέραμε τα βασικά σημεία που μα απασχολούν, ειδικότερα δύο. Ε, το πρώτο από αυτά είναι ότι σε ό,τι αφορά τι αναδιαρθρώσει θέλουμε να υπάρχει μια καλή ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών ε, συμφερόντων, ειδικότερα ανάμεσα στου ε, πίστοτε και του οφειλέτε. Και το δεύτερο σημαντικό σημείο το οποίο αναφέρεται και στο ψηφισμά μας, είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις. Εξετάσαμε λοιπόν, διατρέξαμε όλο το κείμενο σε ό,τι αφορά τα βασικά ζητήματα που μας απασχολούν σε αυτό το τριμερή ε, διάλογο. Περάσαμε και στην κατάρθρο εξέταση και έχουμε τώρα πραγματικά περάσει στην πραγματική εξέταση των ε, ζητημάτων. Θα λάβει ακόμα ένα τρίτο, ε, μια τρίτη συνάντηση και προηγουμένως θα έχουμε ήδη συζητήσει σε τεχνικό επίπεδο περαιτέρω ζητήματα, οπότε αναμένουμε μέσα σε αυτό το τρίτο μερή διάλογο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, τουλάχιστον αυτό φιλοδοξούμε να κάνουμε, έτσι ώστε δηλαδή να υιοθετηθεί η πρόταση υπό την Αυστριακή Προεδρία. Δεν είναι τόσο δύσκολο έτσι κι αυτό το ζήτημα. Απλώ ε, προσπαθούμε συζητώντα παράλληλα διαφορετικά ζητήματα να φτάσουμε στι κατάλληλε λύσεις. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη προσπαθούν από τη δική του πλευρά να διασφαλίσουν όσο περισσότερη ευελιξία μπορούν σε εθνικό επίπεδο, ενώ εμείς από την άλλη πλευρά προσπαθούμε να επιτύχουμε κάποια εναρμόνιση, ώστε να ισχύουν κάποιε βασικέ αρχέ σε ό,τι αφορά τι ε, ε Και προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε εμεί από την πλευρά του Κοινοβουλίου και βέβαια είμαστε στη διάθεση των συναδέλφων για ερωτήματα. Ευχαριστώ. Υπάρχει κανεί που να ζητάει το λόγο. Όχι. Επιτροπή. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω απλώς την ε, εισηγήτρια σε σχέση με την ε, πολύ διεξοδική δουλειά που έχει κάνει σε σχέση με αυτό το φάκελο. Πραγματικά προχωρούμε στους ε, τριμερείς διαλόγους και είμαστε στη διάθεσή σας να σας υποστηρίξουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια κάνετε έτσι ώστε να μπορέσουμε, όπως είπατε και εσείς, να ολοκληρώσουμε τις διαβουλεύσεις πριν από τα τέλη του χρόνου. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, μπορούμε να ολοκληρώσουμε λοιπόν σε αυτή τη φάση την εξέταση του σημείου 28. Μπορούμε να περάσουμε λοιπόν στο σημείο 33, εξέταση δηλαδή σχεδίου γνωμοδότησης ε, σε σχέση με έρευνες που, ε, της ε, Όλαφ σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Ζαμαρή Καβαντά είναι αρμόδιος. Τις παρακαλώ. Είχαμε μια μικρή δυσκολία στο κείμενο και ζήτησα από την κυρία Μαρίν Τελβό να διαβάσει το κείμενο. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που μου κάνετε αυτή την τιμή. Ε, λέει λοιπόν ο κύριος Καβαντά, μετά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τον κανονισμό που διέπει τις έρευνες της Όλαφ έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών. Η Γενική Εισαγγελία θα είναι υπεύθυνη για ποινικέ υποθέσεις και για συνέχεια υποθέσεων ενώπιον των εθνικών δικαστικών αρχών. Η Όλαφ θα είναι αρμόδια για τις ε, διοικητικές έρευνες είναι πιο, έχει πιο περιορισμένες αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελία. Η Επιτροπή θα ήθελε να προβεί σε περιορισμένες αλλαγές για να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών και την καλύτερη αποτελεσματικότητα του έργου της ΟΛΑΦ επικεντρώνεται σε τρία σημεία. Την υποχρέωση της Όλαφ να κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία περιπτώσεις της αρμοδιότητάς της. Δεύτερον, τη μη επικάλυψη των ερευνών και τρίτον, ειδικού ε, κανόνες που θα ισχύουν όπως θα ορίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουν γίνει και ορισμένες ε, τροποποίησεις για την καλύτερη αποτελεσματικότητα του έργου της ΟΛΑΦ. Οι προτάσεις για τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, ανταλλαγή πληροφοριών ως προς το ΦΠΑ, την αρχή του παραδεκτού των αποδεικτικών στοιχείων της ΟΛΑΦ, την καταπολέμηση της απάτης στα κράτη-μέλη και ή τις δραστηριότητες συντονισμού της Όλαφ. Υποστηρίζω αυτές τις τροποποιήσεις, θα ήθελα όμως να εισαγάγω ορισμένες τροπολογίες για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των δύο συμβαλωμένων μερών, τους ενδιαφερόμενους και την τήρηση των ε, αρμοδιοτήτων των δύο οργανισμών, τη συνεργασία των κρατών μελών και την ε, προστασία των καταγγελόντων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε την εκπρόσωπο του κυρίου Καβαντά και ο κύριος ε, Ράντιεφ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Καβαντά, διότι συμφώνησε να αλλάξει την προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών, γιατί με εξέπληξε το χρονοδιάγραμμα. Είμαι σίγουρος ότι πολύ καλή αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί όταν ε, συνεργαστούμε στις τροπολογίες συμβιβασμού. Το κείμενο είναι τεχνικής ε, υφής, αλλά αυτό δεν μειώνει τη σημασία του. Χρειάζεται καλή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και Όλαφ για να προσπιστούν τα ε, χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η Όλαφ δεν θα πρέπει να επικαλύψει την εργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα πρέπει να γιούμε τι γίνεται αν διενεργηθεί έρευνα μεταξύ κράτους ε, που συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλου κράτους το οποίο δεν συμμετάχει. Δεν νομίζω ότι αυτές οι συμφωνίες συνεργασίας αρκούν όταν ε, θέλουμε να αποφύγουμε ενδεχόμενα ε, προβλήματα και κολλήματα του μέλλοντος. Αυτοί είναι τομείς ε, στους οποίους θα υποβάλω τροπολογίες και ελπίζω οι τελικοί συμβιβασμοί να διευκολύνουν την εργασία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Όλαφ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να σχολιάσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Καβαντά γιατί το σχέδιο γνωμοδότησης καλωσορίζουμε την υποστήριξή του στην προσέγγιση μας. Προσπαθούμε να φτάσουμε σημαντικές τροπολογίες για να διασφαλίσουμε τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και επίσης οι τροπολογίες να ισχύσουν από τη στιγμή της λειτουργίας της ΕΠΟ, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι τροπολογίες θα υποβάλουμε ως προς τον κανονισμό της Όλαφ. Και υπάρχουν και περιορισμένες τροπολογίες από τη συνεκτική αξιολόγηση του νομικού πλαισίου που ολοκληρώθηκε πέρσι. Καλωσορίζουμε και την υποστήριξη ως προς τις Γενικές Αρχές Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ΟΛΑΒ. Θα πρέπει να βασιστούμε στην στενή συνεργασία, ανταλλαγή πληροφοριών και συμπληρωματικό χαρακτήρα δράσης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται με ποινικέ υποθέσεις, αλλά η Όλαφ θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη ως προς τις διοικητικές πτυχές προστασίας του προϋπολογισμού και τις χρηματοοικονομικές ανακτήσεις ε, χρημάτων. Θέλουμε λοιπόν να διασφαλίσουμε αυτό το συσχετισμό έτσι ώστε η Όλαφ να μπορέσει να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σε σχέση με αυτό, θα ήθελα να προσθέσω ότι όταν η Όλαφ υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό αφορά την αρμοδιότητα της ΕΠΟ στα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τα μη συμμετέχοντα κράτη όπου η εντολή της Όλαφ θα παραμείνει ως έχει. Και τη στιγμή που υπάρχουν ε, ε, υποψίες ε, εγκληματικών δράσεων, τότε θα περάσουμε αυτές τις πληροφορίες στις εθνικές εισαγγελικές αρχές. Υπάρχουν και τροπολογίες επιτάπητος που αφορούν τη διαφάνεια και συνεργασία μεταξύ των οργανισμών που καταπολεμούν την απάτη και ε, συμβαδίζουν με τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής και θα συνεργαστούμε μαζί σας αν ανακύψουν άλλες τροπολογίες τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ε, θέλει κανένας άλλος να λάβει το λόγο. Η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 22 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Τώρα συνεχίζουμε με το θέμα 34 που είναι η εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Α, είναι ανταλλαγή απόψεων, με συγχωρείτε, για την προστασία των των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρία Μπερζερόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε και τους εκπροσώπους της Κομισιόν και της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και της Γενικής Γραμματείας σήμερα και χαίρομαι γι' αυτό. Ζητώ συγγνώμη, δυσκολεύομαι να μιλήσω, λέει ομιλήτρια. Ε, χαίρομαι γιατί έχω να τους υποβάλω ερωτήσεις και είναι σημαντικό να γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η Γενική Γραμματεία ήδη μου έστειλε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο έλαβα μόλις σήμερα το μεσημέρι και αντικατέστησα μια, ε, ένα συνάδελφο σε μια ψηφοφορία σε μια άλλη επιτροπή. Το ερωτηματολόγιο φυσικά ήταν στα αγγλικά και δεν μπόρεσα να το μελετήσω. Αυτή η αίτηση γνωμοδότηση από την Νομική Επιτροπή θέτει σε ένα εντελώ, εντελώς ε, ιδιαίτερο πλαίσιο, στο πλαίσιο της Cambridge Analytica, κατά την οποία 2,7 ε, εκατομμύρια δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών ε, που ήταν στη διάθεση αυτής της εταιρείας, το οποίο οδήγησε σε χειραγώγηση των των ε, αποτελεσμάτων. Αυτό επιβεβαιώθηκε από το δημοψήφισμα του 2016 για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Αποδεικνύεται ότι κάποια ιδιωτική επιχείρηση μπόρεσε να παραβιάσει βασικούς κανόνες όπως τις προστασίες προσωπικών δεδομένων με σκοπό ε, μια ψηφοφορία που ήταν πάρα πολύ σημαντική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Βρετανία. Η Επιτροπή ασχολείται με την ουσία όπως και η Κομισιόν ΙΜΚΟ. Και με τη γραμματεία συμφωνήσαμε η γνωμοδότηση να σταλεί υπό μορφή επιστολής για να ε, μειωθεί ο χρόνος ε, της διαδικασίας. Τώρα, όσον αφορά το θέμα, η Κομισιόν σκοπεύει να τροποποιήσει του υφιστάμενου κανόνε για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και μάλιστα πριν τι ευρωπαϊκέ εκλογέ, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα να υποβληθούν τροπολογίε σε ε, ε, πρόστιμα σε κόμματα που χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για να επηρεάσουν τι εκλογέ. Επίση, θέλει να κινηθεί κατά του διαδικτυακού χειρισμού των ε, εκλογέων και των χειρισμών με πολιτικούς σκοπούς. Ε, το θέμα είναι κατεπήγον ε, και αφορά τη διαφήμιση, την κυβερνοασφάλεια, την προστασία των, των ε, ε, προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων ψηφοφόρων και την ελευθερία της γνώμης τους, επηρεάζει τη δημοκρατία και μια σειρά από άλλα θέματα. Επίσης, πρέπει οι κανόνες να είναι αυστηροί και η ταχύτητα δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε βιαστικές λύσεις πρέπει βραχυπρόθεσμα ε, ε, να ασχοληθούμε και με τα ευρωπαϊκά αλλά και με τα εθνικά πολιτικά κόμματα. Μια σειρά από γνωμοδοτήσεις έχουν σχέση με τις ε, διαδικτυακές εκλογικές και διαφημιστικές εκστρατείες, όπως επίσης και με τη στόχευση συγκεκριμένων ομάδων εκλογέων. Υπάρχει ένας κίνδυνος να πέσουμε ε, σε ένα είδος ε, αστυνομικής καρικατούρας παντός ελέγχου. Δεν θα πρέπει να παραβιαστούν τα δικαιώματα των πολιτικών κομμάτων της Ευρώπης που δεν θα πρέπει να θέσουμε κανόνες που να είναι πολιτικά ορθοί ή ευρωσυμβατοί. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Κομισιόν θέλει να δημιουργήσει ένα νέο, ε, μια νέα μορφή οικονομικών ε, προστήμων με βάση το άρθρο 27 για όποιον θέλει να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές εκλογές. Για μένα υπάρχει ένας κίνδυνος. Είναι σημειολογικός, αλλά ε, με ενδιαφέρει το νόημα των λέξεων. Ποιος θα το κρίνει αυτό. Μια αρχή μας λέει η Κομισιόν, που θα αποτελείται από εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Δεν, δεν εξασφαλίζεται η ε, διαδικασία εδώ. Δεν υπάρχουν διαδικαστικές εγγύησεις. Τα κόμματα, ε, εγώ δεν είμαι ευρωσκεπτικίστρια, κάποιοι από εμά είναι, πιστεύω ότι έχουν δικαίωμα να είναι και αυτό είναι δημοκρατικό δικαίωμα. Δεν μπορεί να καταδικαστούν μόνο και μόνο γι' αυτό. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ε, μιλήσουμε για το θέμα αυτό που είναι και πολιτικό και νομικό. Ευχαριστώ κύριο Ραντεφ, λέει ο πρόεδρος. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το θέμα των προσ... της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ιδίως όταν αυτά αφορούν τις δημοκρατικές ευρωεκλογέ είναι πολύ σημαντικό. Είναι κρίσιμη σημασία, θα έλεγα. Οι εξελίξεις της επιγραμμικής επικοινωνίας τα τελευταία χρόνια επιτρέπουν αλληλεπίδραση μεταξύ πολιτικών και πολιτών, η οποία να είναι όλο και πιο ε, σαφής και ε, εκ του σύνεγγης. Και αυτό φυσικά αυξάνει τους κινδύνους των παράνομων, της παράνομης επεξεργασίας των στοιχείων των πολιτών. Δυστυχώς πριν από λίγους μόνο συνέβη αυτό και ήμασταν μάρτυρες του τρόπου με τον οποίο πάνω από 50 εκατομμύρια άνθρω... Ε, δεδομένα πάνω από 50 εκατομμυρίων ανθρώπων ε, χρησιμοποιήθηκαν, μερικά από τα οποία και για πολιτικούς σκοπούς κατά την εκλογική εκστρατεία του Προέδρου Τραμπ και στην εκστρατεία για το δημοψήφισμα για το Brexit. Η κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων και των κανόνων προστασίας τους μπορεί να επηρεάσει τη δημοκρατική συζήτηση και τη δημοκρατία και αυτό μπορεί να επηρεάσει τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές για το Κοινοβούλιο. Αυτό δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε. Παρότι ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο GDPR, ε, ετέθη ενισχύει από φέτος το Μάιο, οι κανόνες δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική πρόληψη και την εισαγωγή κυρώσεων στις περιπτώσεις κατάχρησης των προσωπικών δεδομένων, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν τις ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές με σκοπό την εξασφάλιση της δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών αξιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε, προετοίμασε την ε, υπομελέτη πρόταση που προτείνει την επιβολή κυρώσεων σε ευρωπαϊκά ε, κόμματα και οργανώσεις που παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων όταν υπάρχει διαμφισβήτητη απόδειξη ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για σκόπιμη επιρροή ή ε, προσπάθεια επιρροής του αποτελέσματος των εκλογών. Είναι λοιπόν σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι αυτές οι κυρώσεις θα επιβάλλονται όχι μόνο σε πολιτικά κόμματα και ιδρύματα, αλλά και σε άλλα άτομα και οργανισμούς, εάν αποδειχθεί ότι με τις πράξεις τους σκοπίμως επηρέασαν ή επεχείρησαν να ε, επηρεάσουν το αποτέλεσμα ε, ε, υπέρ ενός πολιτικού κόμματος οι προτινόμενες αλλαγές σκοπό έχουν να ενισχύσουν το έργο της ε, Αρχής Προστασίας ε, ε, Προσωπικών Δεδομένων με την δημιουργία ελέγχων και να επιβάλλουν στοχευμένες κυρώσεις σε πολιτικά κόμματα και ιδρύματα, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, εάν αποδειχθεί ότι έχουν παραβιάσει τα προσωπικά δεδομένα, όταν υπάρχει ξεκάθαρη απόδειξη ότι έχουν επηρεάσει ή έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Η πρόταση που υποβλήθηκε σχετικά είναι κατά τη γνώμη μου ορθή. Ε, ανησυχώ λίγο για τις ε, προθεσμίες για, τα, για τους ελέγχους, τα check-up. Δεδομένου της ουσία, της ουσίας, τα check-up αυτά θα πρέπει να γίνονται γρήγορα ώστε όταν αποκαλύπτεται ότι έχουν ε, γίνει παράνομες πράξεις να σταματήσουν και οι υπεύθυνοι να υφίστανται κυρώσεις χωρίς αυτό να επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη συνεργασία μας επί του θέματος. Είναι σημαντικό να δουλέψουμε γρήγορα ώστε οι προτάσεις να τεθούν εν πριν από τις επερχόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Nous abordons ένα σημαντικό θέμα, γιατί ε, ε, και η Cambridge Analytica μας έδειξε πως έχει κατάσταση το δημοψήφισμα του 16 για το Brexit επηρεάστηκε από τη χρήση ορισμένων προσωπικών δεδομένων. Και φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στις ευρωεκλογέ. Καλά, φυσικά κανένας δεν το θέλει αυτό. Από αυτά τα ευγενή αισθήματα βέβαια το... φτάνουμε σε ένα κείμενο που είναι πολύ κατασταλτικό. Μιλάμε για κυρώσεις στα κόμματα, στους οργανισμούς, στα ιδρύματα που θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν προσωπικά δεδομένα για πολιτικούς λόγους. Εδώ δέχομαι τις προβλέψεις ε, της εισηγήτριας. Δηλαδή υπάρχουν πολύ καλά αισθήματα και προθέσεις, αλλά φτάνουμε σε μία αστυνομική δομή, μία ε, δομή αστυνόμευσης. Εγώ δεν έχω αυταπάτες βεβαίως, είμαι μέλος ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος που εσείς θα το, θα το θεωρούσατε ότι υποστηρίζει τους ευρωσκεπτικιστές. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό, αλλά ας το δεχθούμε σαν υπόθεση εργασίας. Αυτή η μεμψημυρία και η, ε, ο λεπτομερής έλεγχος οδηγεί στον ευρωσκεπτικισμό γιατί δεν υπάρχει ίση μεταχείριση και αυτό θα αφορά και το, τη δική σας διαδικασία ελέγχου. Δύο παραδείγματα. Μιλάμε για κυρώσεις όχι μόνο κατά των κομμάτων, αλλά και αυτών που θα προσπαθούσαν να επηρεάσουν. Τι σημαίνει αρχίζουμε να προπυλακίζουμε τους ανθρώπους και γίνεται λόγος για μία επιτροπή ανεξάρτητων προσωπικότητων ε, για την εξέταση του στήματος. Μα εδώ θα περιλάβετε και τους ευρωσκεπτικιστές, δεν νομίζω. Δηλαδή κινούμαστε προς τη λογική του Orwell με το έργο του 1984. Ε, θα έχουμε μια κοινωνία όπου ο μεγάλος αδελφός ε, βρίσκεται από πάνω. Κύριε Λεμπρετόν, υπάρχουν πολιτικά κόμματα στην ε, Ευρώπη και στη Γαλλία που πληρώνονται από το μεγάλο αδελφό. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός. Και εδώ εντάσσεται ακριβώς και αυτό που αναφέρατε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι από τη Γενική Διεύθυνση Just και σε σχέση με αυτό το πακέτο θα ήθελα να επαναλάβω τα πλαίσια ε, αυτού του πακέτου. Τα συμφραζόμενα αφορούν τον κίνδυνο που μπορεί να πλήξει τις ευρωεκλογές και αυτό το είδαμε μετά τη δράση της ε, Cambridge Analytica που ε, άρπαξε στοιχεία από το Facebook. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το νομοθετικό σκέλος και το μη νομοθετικό. Ε, το μη νομοθετικό αφορά την επικοινωνία, την παρουσίαση αυτού του πακέτου για την εξασφάλιση των δίκαιων ελεύθερων εκλογών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε και ε, γενική, γενικές κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι κατευθυντήριες γραμμές ε, μετά από την έγκριση του κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα, έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές τα κόμματα και τα εμπλεκόμενα μέρη να ασχοληθούν με την ε, προστασία δεδομένων. Αυτό αφορά το μη νομοθετικό σκέλος. Υπάρχει και μία σύσταση προς τα κράτη-μέλη και τις αρχές τους και τα πολιτικά κόμματα, η οποία αναγνωρίζει όπως και η συνθήκη τη σημασία των ε, πολιτικών κομμάτων για την ε, ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι τα δομικά στοιχεία. Θα ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με βάση τους προϋπάρχοντες κανόνες για την ε, προστασία δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές, οι αρχές ε, προστασίας του κυβερνοχώρου για την ακαιρεότητα των εκλογών και θα υπάρχει ένα ε, συναφές ευρωπαϊκό δίκτυο που συμβαδίζει με τον ε, νόμο. Επίσης, προώθηση της διαφάνειας στην πολιτική ζωή, όπου ζητάμε τα παρκάτη μέλη να υποστηρίξουν τη διαφάνεια και τα πολιτικά κόμματα να έχουν διαφάνεια ως προς τη διαφήμιση και χρηματοδότησή τους. Υπάρχει και ένα τρίτο, ένας τρίτος πυλώνας που αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με βάση τις πρακτικές που υπάρχουν για να εξασφαλίσουμε την, τον κυβερνοχώρο και υπάρχει και μία νομική πρόταση Ε, στην περίπτωση παραβίασης ε, προσωπικών δεδομένων για ε, να επηρεάσει κανείς το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν τις κατάλληλες κυρώσεις γιατί αυτό σημαίνει ότι προσπαθεί να υπάρξει επιρροή για το εκλογικό αποτέλεσμα. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν και ένα άλλο συμβαλόμενο μέρος για την προστασία δεδομένων και θα ήθελα να δώσω το λόγο σε, στο συνάδελφο για να μας μιλήσει για θέματα νομικής βλάβης. Τι συνάδελφο. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση γιατί εξετάσατε την πρότασή μας εμείς προτείνουμε μία στοχοθετημένη τροποποίηση ως προς το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Θέλουμε να δράσουμε εκεί που μπορούμε, εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητες για την περίπτωση παραβίασης πολιτικών δεδομένων, προσωπικών συγγνώμη δεδομένων από τα πολιτικά κόμματα. Γιατί μιλάμε για τα ευρωπαϊκά κόμματα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δυνατότητα δράσης μέσω του νομικού αυτού μέσου. Μιλάμε για εφαρμογή ενός μηχανισμού που κινεί από την αρχή, ε, από την αρχή της προστασίας δεδομένων και ε, δεν μπορεί κανείς να βασιστεί σε καταγγελίες απλώς που είναι ασύστατες, άρθρα εφημερίδων, κουτσομπολιά και τέτοια. Θέλουμε να επιβάλλονται κυρώσεις με βάση ε, την Επιτροπή Ανεξάρτητων ε, Εμπειρογνωμόνων η οποία θα έχει συσταθεί και θα παρτίζεται από έξι πρόσωπα, ε, δηλαδή από τα τρία θεσμικά όργανα, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή. Θα είναι χρηματικές ε, οι κυρώσεις και βεβαίως υπάρχει και το θέμα της χρηματικής κύρωσης 5% του προϋπολογισμού καθώς και την απαγόρευση συμμετοχής στη χρηματοδότηση του επόμενου έτους. Εάν υπάρχει, λοιπόν, βάση, αν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία για την επιρροή ε, του εκλογικού αποτελέσματος. Αναμένουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής σας στην πρόταση, θα την ε, μελετήσουμε και έχουμε διάλογο με τις Επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΑΦΚΟ και θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσει τάχιστα επί του θέματος γιατί θα θέλαμε να προτρέξουμε τον, εκλο... ευρωεκλογών του 2019 και ίσως ο συνάδελφος για την προστασία δεδομένων θα μπορούσε να λάβει το λόγο. Merci. Je vais répondre en français puisque la plupart... Θα απαντήσω στα γαλλικά γιατί οι περισσότεροι παρεμβαίνοντες είναι Γάλλοι. Σε σχέση τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για την προστασία προσωπικών δεδομένων, θεωρώ ότι αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ένα στόχο να μπορέσουν τα εμπλεκόμενα μέρη στην εκλογική διαδικασία να υποστηρίξουν τους βασικότερους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων διότι είδαμε ότι πολλά συμβαλόμενα μέρη, είτε πολιτικά κόμματα, είτε εταιρείε συλλογής δεδομένων και ανάλυσης δεδομένων, κοινωνικά δίκτυα και ούτω καθεξής, δεν εφαρμόζουν πάντα τους κανόνες που ισχύουν από το Μάιο. Έτσι, έτσι ε, διασαφηνίζονται τα δεδομένα και θα έχουμε την πρώτη εκλογική αναμέτρηση δυνάμει αυτών των κανόνων, γι' αυτό τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να ξέρουν πιο σημαντικούς κανόνες. Έχουμε ένα έγγραφο που πιστεύουμε ότι είναι ε, αρκετά σαφές, έχουμε ένα checklist για να δούμε κατά πόσο τα πολιτικά κόμματα έχουν συλλέξει προσωπικά δεδομένα, αν ναι, για ποιο λόγο. Θα πρέπει κανείς να προσέξει αυτά τα δεδομένα. Θα πρέπει να ελέγξουν την εταιρεία προέλευσης για την εξέταση αυτών των δεδομένων. Δεν λέμε ότι τα πολιτικά χρώματα, κόμματα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα, γιατί στόχος των πολιτικών κομμάτων είναι να περάσουν ένα μήνυμα, αλλά θα πρέπει να γίνει νόμιμα. Πολλοί αναφέρθηκαν στην Cambridge Analytica, περίπτωση που ίσχυε πριν τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και θα πρέπει να το υπενθυμίσουμε και για τις προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου θα πρέπει να υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές προστασίας δεδομένων. Και οι αρχές αυτές διαπίστωσαν ότι υπήρξε παραβίαση προστασίας των προσωπικών αυτών δεδομένων. Δεν μιλάμε για κόμματα υπέρ της Ευρώπης ή ευροσκεπτικιστές. Έγινε παραβίαση της νομοθεσίας. Και από αυτό το σημείο εκκίνησης θα δει αυτή η αρχή κατά πόσο αυτή η παραβίαση προστασίας έγινε με στόχο επιρροής του τελικού εκλογικού αποτελέσματος. Στην περίπτωση της Cambridge Analytica, η έρευνα που δεν διενεργήθηκε από την ICO, την αρμόδια Βρετανική Αρχή, έδειξε σαφέστατα τα αποτελέσματα της έρευνας, όμως που να έχουμε περιπτώσεις όπου ένα συμβαλόμενο μέρος έκανε ένα λάθος. Δεν προστάτευσε τα δεδομένα, του επιβλήθηκαν κυρώσεις βάσει νόμου, αλλά δεν ήθελε να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Άρα δεν θα υπάρχουν επιπρόσθετες κυρώσεις. Αυτό θέλαμε να υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Well. So, thereby... ε, σας ευχαριστώ και εγώ. Τώρα μπορούμε να, στα, να, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση επί του 34, να περάσουμε στο 35, σημείο 35, που αφορά τη συζήτηση της ασφάλισης αστικής ευθύνη για τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων κλπ. Για μία ακόμα φορά η κυρία Μπερζερό είναι η συγγήτρια. Ξέρω, παίρνω και πάλι το λόγο για ένα θέμα που είναι καυτό. Θα παρουσιάσω εν συντομία την νομική μου θέση για την πρόταση οδηγίας που τροπολογία που τροποποιείται είναι η οδηγία της 7 Δεκεμβρίου 2009 που αφορά την ασφάλιση αστικής ευθύνης για τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων και την επιβολή της υποχρέωσης ασφάλισης για τέτοια ευθύνη. Η πρόταση οδηγίας έχει σκοπό να αντιποκριθεί στις νέες απαιτήσεις προστασίας θυμάτων, ροδικών ατυχημάτων σε χώρους πέραν από τους χώρους κατοικία της ή όταν ο οδηγός που προκαλεί προέρχεται από άλλο κράτος μέλος. Μετά την, η οδηγία του 2009 καθιστά την ασφαλιστική ευθύνη για τη χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων προ, ε, υποχρεωτική έχουν εμφανιστεί διάφορες δυσκολίες. Η Κομισιόν λοιπόν αναγκάστηκε να διαπιστώσει ότι πρέπει να προσαρμοστούν κάποια σημεία για την επίτευξη του βασικού στόχου που είναι η προστασία των ε, θυμάτων των ε, οδικών ατυχημάτων σε διασυνοριακές περιοχές. Σκοπός είναι να τροποποιηθεί η οδηγία του 2009 επί πέντε ε, θεμάτων που είναι ουσιαστικά. Το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας είναι το άρθρο 1 της οδηγίας του 2009 ο έλεγχος της ασφάλισης για να μην οδηγούν χωρίς ασφάλειες, άρθρο 4, η εναρμόνιση και η αναθεώρηση των ελάχιστων ποσών κάλυψης, άρθρο 9 της οδηγίας του 2009, η περίπτωση της αφαιρεγγιότητας του ασφαλιστή ε, και η τροποποίηση και η ανάληψη ευθύνης ε, για το δικόγραφο αγωγής. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι η πρόταση αυτή διορθώνει τα θέματα πρακτικά και νομικά της Οδηγίας 2009. Όσον αφορά τον έλεγχο ασφάλισης, είναι σημαντικό να υπάρξει απαγόρευση της αρχής των να ελέγχουν τα κράτη-μέλη την αστική ευθύνη των ε, οχημάτων που συνήθως βρίσκονται στο εδαφός από ένα κράτος μέλος ή των τρίτων χωρών που εισέρχεται στο εδαφός τους. Ε, ε, ε, να επιτρέπεται να κάνουν μη, καταχρηστικές, μη καταχρηστικούς ελέγχους. Δηλαδή, μέσω τεχνικών που δεν, δεν επιβάλλουν την, το σταμάτημα του αυτοκινήτου με από τις, τους αριθμούς κυκλοφορίας να μην επιβάλλονται διακρίσεις και με αναλογικό τρόπο. Αυτό επιτρέπει να μπορεί κανείς να, ε, μην, να μην επιτρέπει την οδήγηση χωρίς ασφάλιση. Όσον αφορά την κάλυψη ε, για ηλική σωματική βλάβη, υπάρχει αυτή η νέα πρόταση όπου τα κράτη μπορούν να ξεπεράσουν το ελάχιστο και το ποσό αυτό θα αναθεωρείται κάθε πενταετία, λαμβάνοντας υπόψη την, τις τιμές. Όσον αφορά Λέω ό,τι θέλω, λέει, λέει η ομιλήτρια, με συγχωρείτε. Λοιπόν, όσον αφορά ε, τα ατυχήματα, η πιθανότητα αποζημίωσης ε, είναι μακαροσκελής και σύνθετη και θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ταχείας καταβολής της αποζημίωσης στα θύματα. Σε, τέλος, η πρόταση που περιλαμβάνει τη δημιουργία σε κάθε κράτος μέλος ε, ένα ταμείο οικονομικής αποζημίωσης από τις εθνικές αρχές όσον για την περίπτωση της, ε, του μη φερέγγιου ασφαλιστή. Σε περίπτωση που το θύμα βρίσκεται σε ένα κράτος όταν δεν πρέπει να αναλαμβάνεται ευθύνη για την περίπτωση της, του αφαιρέγγιου ασφαλιστή. Επίσης, πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να διευρυνθεί σε όλα τα κράτη και αυτό για μένα είναι πρόοδος. Επίσης πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάληψη των περιπτώσεων αυτών ε, από τον ίδιο τρόπο από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από οποιοδήποτε και είναι το κράτος μέλος και αυτό με βρίσκει σύμφωνη. Ο στόχος είναι ουσιαστικά να υπάρχουν λιγότερες ασφαλιστικές απάτες, περισσότερη διαφάνεια με τον ε, εντοπισμό της δήλωσης του ή του δικογράφου αγωγή. Τώρα, όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή οδηγία, οδηγίας, ε, αντιλαμβάνομαι και συμμερίζομαι την ε, επιθυμία την, να ληφθεί υπόψη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την κυκλοφορία οχημάτων. Όμως θεωρώ ότι ο ορισμός είναι εξαιρετικά περιοριστικός και μπορεί να εξαιρούνται κάποια οχήματα τα οποία συνήθως δεν έχουν σκοπό να ε, αποτελούν οχήματα μεταφορά, αλλά που ενδεχομένως προκαλούν ατυχήματα και την προηγούμενη φορά με ρωτήσατε από αυτού. Ας πούμε τα, τα ε, τα πατίνια που, είναι, που έχουν γεμίσει τα πεζοδρόμια του Παρισιού. Και υπάρχουν οχήματα ε, που εμπίπτουν σε αυτή την αγωγία. Τα οχήματα που κυκλοφορούν και χρησιμοποιούνται ε, για την κατασκευή δημοσίων έργων σε διαμεθοριακά μπορούν και αυτά να προκαλέσουν ατύχημα. Θεωρώ ότι ο ορισμός της κυκλοφορίας του οχήματος θα πρέπει να είναι ο αυρύτερος δυνατόν ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή προστασία στα θύματα των ατυχημάτων. Υπό την έννοια αυτή κατέθεσα τροπολογία από αυτού. Ε, φυσικά περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας και πρέπει να διευκρινίσω ότι η προθεσμία υποβολής ε, τροπολογιών είχε ε, οριστεί για σήμερα το μεσημέρι. λίγο, είναι λίγο σύντομη γιατί είμαστε σήμερα στις 5 και και έτσι μάλλον πρέπει να μετατεθεί για τις 22. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Uh-huh. Uh if um, Madame Bergeron would, like uh, that, we can... Εάν uh, το θέλει η κυρία Μπερζερόν, μπορούμε να έχουμε νέα προθεσμία 22, 22 Νοεμβρίου στις 6 no problem with that. Δεν υπάρχει πρόβλημα από ό,τι βλέπω από αυτού. Μπορούμε λοιπόν να ανακοινώσουμε αυτή την προθεσμία, γιατί το να έχει λήξει ήδη η προθεσμία είναι ασυνήθιστο. Κύριο Βόγκεν, ευχαριστώ. Επί της αρχής χαιρετίζω αυτή την τροποποίηση της οδηγίας που προτείνει η Επιτροπή και μπορώ να υποστηρίξω για τις τροπολογίες της συγκήτριας. Ωστόσο, εγώ θα υποβάλω εμ, κάποιες τροπολογίες ό,τι αφορά τρία-τέσσερα σημεία για να αλλάξουν. Καταρχήν χαιρετίζω και εγώ το γεγονός ότι υπάρχει καταρχήν ένα ελάχιστο ποσό κάλυψης ε, σε ό,τι αφορά σε εναντί προσώπων ε, και το οποίο ποσό βρίσκεται πάνω από το ε, μέσο του μίσεως των κρατών μελών, αλλά αλλά θεωρώ πως αυτό το ποσό των 6.600 ευρώ είναι πολύ χαμηλό. 6 ε, εκατομμυρίων, συγγνώμη, 600.000 και θα έπρεπε να πάει στα 10 εκατομμύρια. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά ε, τα νέα είδη οχημάτων, αυτά τα segways, τα ηλεκτρικά πατίνια ή άλλα ηλεκτροκίνητα τέτοια μικροοχήματα, μπορεί προφανώ η χρήση αυτή αυξημένη του να οδηγήσει και σε περισσότερα ατυχήματα και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει κατάλληλη προστασία και η γρήγορη εκταμείευση των αποσημειώσεων σε αυτέ τι περιπτώσει. Ωστόσο, τίθεται το ζήτημα τη συγκρισιμότητα αυτών των νέων οχημάτων. Δηλαδή θα πρέπει καταρχήν να τα εντάξουμε σε μια κατηγορία. Είναι περισσότερο μοτοσυκλέτε, α πούμε ή περισσότερο ποδήλατα. Μετά η μεγαλύτερη διάθεση δημόσιων χώρων με λιγότερα οχήματα ε, και τα ζητήματα βέβαια που μας απασχολούν σε ό,τι αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανσης πρόκειται για ζητήματα τα όλα αυτά μας απασχολούν και ακριβώς δεν θέλουμε για αυτόν τον λόγο να δημιουργήσουμε με αυτή τη νέα οδηγία προβλήματα για αυτούς τους νέους τύπους οχημάτων. Πάντως, με την οδηγία θα επιβάλλεται υποχρεωτικά για τα κράτη-μέλη η θέσπιση ορισμένων κανόνων. Επίσης, σε ό,τι αφορά κάποιες στοιχείες προστασίας των καταναλωτών, να πω ότι θεωρώ ως ενδεδειγμένο να υπάρξει η θέσπιση ενός συστήματος bonus μάλους ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τον υπολογισμό των ασφαλίστρων ε, και βέβαια το σύστημα του υπολογισμού του bonus μάλους θα πρέπει να είναι διαφανές. Τέλος, ε, σε ό,τι αφορά την μελλοντική τεχνολογική εξέλιξη θα πρέπει στην αξιολόγηση αντικτύπου να αναφέρεται ε, πως ε, η υποχρεωτική ε, ασφάλιση, αστική ασφάλιση για τα οχήματα θα ισχύσει και θα πρέπει να ισχύσει και για τα ημιαυτόματα και αυτόματα οχήματα γιατί βέβαια ο στόχος είναι να υπάρχει πάντοτε η προστασία και η αποζημίωση για τα θύματα τέτοιων οχημάτων, αυτονόμων δηλαδή και μη αυτονόμων αυτοκινήτων. Ένας αριθμός ατυχημάτων που ήδη έχουν λάβει ε, χώρα καταδεικνύει ακριβώς ότι θα πρέπει να υφίσταται η προστασία των ευρωπαϊκών πολιτών έναντι τέτοιων ε, ατυχημάτων. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει, και εδώ το αναφέρω ειδικότερα στο άρθρο 28C, ε, μια ιδιαίτερη ε, ε, μελέτη αυτού του ζητήματο και υποχρεωτική διάταξη σε ό,τι αφορά την ασφάλιση αυτών των οχημάτων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Η Επιτροπή θέλει να σχολιάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Θα ήθελα καταρχήν να σε ευχαριστήσω και πάλι σε ό,τι αφορά τη θετική προσέγγιση της ε, δική σας πρόταση σε ό,τι αφορά δηλαδή τις τροπολογίες που προτίθεται να υποβάλει. Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογής και το ότι δηλαδή είναι υπερβολικά περιοριστικό, αν θέλετε, το πεδίο εφαρμογή. Εμεί δεν θέλουμε να υπαραχωρήσουμε σε αυτή τη φάση από τη δική μα πρόταση. Πάντω, η προστασία των θυμάτων ε, ήταν το, το, το, ο απότερο στόχο, αν θέλετε, η βασική μα αρχή ε, στο νου μα από την πλευρά τη DG όταν ε, προετοιμάζαμε αυτή την ε, πρόταση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες ανησυχίες που εκφράστηκαν, να πω ότι λάβαμε κάποια σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης ότι τα ελάχιστα ποσά κάλυψης της ασφάλισης θα πρέπει να αυξηθούν αλλά δεν έχουμε κάποια δεδομένα στη διάθεσή μας και γνωρίζετε ποια είναι η θέση της Επιτροπής. Δηλαδή οτιδήποτε προτείνουμε θα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία και το μόνο που μπορούσαμε να προτείνουμε αξιολόγηση αντικτύπου, όχι κάτι παραπάνω. Πάντως τα ελάχιστα αυτά ποσά κάλυψης ισχύουν μόνο σε χώρες καταστάσεις και στα σχετικά θέματα των θυμάτων, δηλαδή στο πλαίσιο της τέταρτης αλλά δεν ισχύουν, για παράδειγμα, αυτές οι διατάξεις σε ό,τι αφορά το σύστημα της πράσινης κάρτας. Σε εκείνες τις περιπτώσεις ε, ισχύει πάντοτε το υψηλότερο ποσό από εκείνα που μπορούν να ισχύσουν, δηλαδή στο πλαίσιο μια διασυνοριακή κατάσταση. σε αυτέ τι περιπτώσει, λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ύψο τη αποζημίωση, ισχύει το υψηλότερο όριο. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά τα νέα αυτά οχήματα που εμφανίζονται στου δρόμου, είναι δύσκολο πραγματικά να πούμε κατά πόσο ένα ηλεκτροκίνητο ποδήλατο θα πρέπει να θεωρείται ένα είδος ε, μοτοσυκλέτας, ε, μοτοσακού ή οτιδήποτε άλλο και πάλι εδώ δεν είχαμε δεδομένα στη διάθεσή μας για να καταδείξουμε ότι για παράδειγμα τέτοιου είδου ηλεκτροκίνητα ποδήλατα είναι πιο ασφαλή από μοτοσακό ή οτιδήποτε άλλο. Και από την πλευρά του θύματο, βέβαια, δεν παίζει κανένα ρόλο αν τελικά ε, εκείνο που τον χτύπησε είναι ε, ένα ηλεκτροκίνητο ποδήλατο ή ένα ε, εντό μοτοσυκλέτας ή οτιδήποτε άλλο. και δεν έχει κανένα νόημα να προβλέπουμε κάτι εδώ και από την άλλη πλευρά να ακούμε στην Επιτροπή Αναφορών, για παράδειγμα, από την πλευρά των θυμάτων ή των συγγενών, ότι θα πρέπει η Επιτροπή να αναλάβει περισσότερη δράση γιατί η προστασία που παρέχεται αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκής. Άρα λοιπόν η θέση μας ήταν ότι πάντοτε σεβόμενη την αρχή της επικορικότητας, τα κράτη-μέλη προφανώς μπορούν να Εξαιρέσουν ορισμένου τύπου οχήματο από το Ταμείο Εγγύσεων, ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε και θεωρούμε ότι προσφέρουμε την κατάλληλη λύση, μια, μια σωστή λύση. Γιατί ε, προφανώς ο, εάν ο βαθμός κινδύνου ενός ε, τέτοιου οχήματο είναι χαμηλό, τότε δεν υπάρχει κίνδυνο σε ό,τι αφορά το Ταμείο Εγγυήσεων. Ενώ, εάν από την άλλη πλευρά έχουμε για παράδειγμα ένα όχημα το οποίο έχει ψηλότερο κίνδυνο και κατά συνέπεια σε κίνδυνο βρίσκονται υψηλά κονδύλια, για να είμαι λίγο κοινικό, τότε χρειαζόμαστε ακριβώ ένα τέτοιο ταμείο. Επίση, θεωρούμε πω ε, τα ασφάλιστα σε αυτέ τι περιπτώσει θα είναι αντίστοιχα ακριβώ, θα ανταποκρίνονται στον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει το κάθε όχημα. Με το ποδήλατο δηλαδή δεν μπορεί κανείς να προκαλέσει για παράδειγμα ένα ε, μείζον συνδρομικό ατύχημα στην, σε μια περίπτωση δηλαδή το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι ε, ε, ένα άτομο να τραυματιστεί από το τρένο. Άρα λοιπόν το ασφάλιστρο ανταποκρίνεται στο βαθμό κινδύνου. Το ασφάλιστρο όπως αυτό υπολογίζεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Αλλά γνωρίζουμε βέβαια ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις δεν ε, ενδιαφέρονται πολύ να ασφαλίσουν αυτά τα νέα οχήματα γιατί γενικά η ασφάλιση αυτή η διαστικής ευθύνη δεν είναι πολύ προστατοφόρα για αυτές τις επιχειρήσεις αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή αυτή είναι η λύση και η εξαίρεση ορισμένων τύπων οχημάτων πάντοτε ήταν κάτι που αποφεύγαμε στην οδηγία ε, το αφήναμε δηλαδή στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών, ώστε να μην υπάρξει υπερβολική περιπλοκότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί βέβαια είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθούμε όλα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο τεχνολογικών εξελίξεων στον ε, ε, τομέα των οχημάτων. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αυτόνομα και αυτόνομα οχήματα, η δική μας θέση είναι ότι η οδηγία ήδη τα καλύπτει και αυτό καταρχήν είναι βασική μας τοποθέτηση σε οποιαδήποτε περίπτωση ατυχήματος, δηλαδή καλύπτονται ήδη. Παρότι βέβαια ε, σε αυτές τις περιπτώσεις η... το ατύχημα προκαλείται από την τεχνολογία που έχει ένα άτομο. Αλλά παρόλα αυτά σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υφίσταται η αστική ευθύνη για την αποζημίωση και από εκεί και μετά βέβαια υπάρχουν όλα τα περαιτέρω ζητήματα όπως η αξιοπιστία του προϊόντος ή για παράδειγμα μπορεί κανείς να ασκήσει αγωγή κατά του κατόχου της υποδομής, δηλαδή του ίδιου του, του, κατασκευαστή του οχήματο και ούτω καθεξής. Ε, πάντως θεωρούμε ότι σε ό,τι αφορά αυτό το τύπο οχήματο ε, η οδηγία είναι επαρκής και απλώς ενδεχομένω να χρειάζεται να προσθέσουμε μια περαιτέρω διευκρίνηση σε μια τελογική σκέψη ή κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους ε, πολύ και α, ε, α, αυτά από τη δική μου πλευρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κι εγώ. Οπότε μοιάζει ότι το θέμα αυτό μπορεί να το ολοκληρώσουμε. να Τελειώσουμε με το 35 και να πάμε στο πιθανότατα τελευταίο θέμα της σημερινής συνεδρίασης, το 36, ε, εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για τη θέσπιση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Λεμπρετόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη δεν είναι απλώς ε, η Ήπειρος, είναι και ο πολιτισμός που ξεκινά από τον ε, ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και έχει επηρεαστεί από τον χριστιανισμό. Γι' αυτό η Ευρώπη δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα οικονομικό οικοδόμημα, πρέπει κυρίως να δώσει αξία τον πολιτισμό των κρατών μελών της για να προωθήσει τον πλούτο και την πολυμορφία αυτού του, πολιτισμού. Για τον λόγο αυτό το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και το άρθρο 5 της Συνθήκης για την ε, ίδρυση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει επίσης την πρόθεση της κοινή πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπάρχει το, το πρόγραμμα ε, Δημιουργική Ευρώπη από το 1921 στο 1927 που ε, είναι αρκετά περιστασιακό. Το πρώτο σκέλος το 2014 ήταν ο πολιτισμός μέσα ενημέρωση και διατομεακό σκέλος. Είναι, είναι φυσιολογικό η Νομική Επιτροπή να συνεισφέρει στην ανανέωση του ωραίου αυτού έργου και υπό την έννοια αυτή σας προτείνω κάποιες τροπολογίες. Ε, φαινομενικά είναι πολλές ε, γιατί είμαι ε, λίγο προσεκτικό στις λεπτομέρειες. Όταν βλέπω ένα κείμενο προσπαθώ να το βελτιώσω, αλλά δεν πρόκειται για πολύ βαθιές τροποποίησεις, επειδή το κείμενο είναι αρκετά καλά στημένο. Η πιο ενδιαφέρουσα τροπολογία για την Επιτροπή μας είναι αυτή που αναφέρει την ανάγκη να δοθεί αποτελεσματική προστασία στην πνευματική προστασία. Γιατί στο κείμενο περιέργως δεν γίνεται μεγάλη αναφορά. Είναι ένα κείμενο που αφορά τα οπτικοακουστικά και φυσικά υπάρχει και εδώ ανάγκη για ιδιαίτερη προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων και των δημιουργών και το θέμα ε, δεν πρέπει να περιοριστεί σε ε, οικονομική βοήθεια. Έχει, υπάρχει μεγάλη πόλωση, χρειάζεται και επαρκής ε, νομική προστασία των έργων και των δημιουργών τους. Έτσι έχουμε τροπολογία 5 και 16 που διώκει τη σύνδεση με άλλα κείμενα που ήδη ψηφίσαμε. Η, κατά την άποψή μου, οι, αυτές είναι οι βασικές αλλαγές που προτείνω. Είναι συμπληρώματα θα έλεγα παρά αλλαγές αυτές καθευτές. Κατά τα λοιπά υπάρχουν κάποιες εκφράσεις που θεωρώ ότι είναι αδέξιες και θα ήθελα να διορθωθούν. Επανειλημμένως αναφέρεται ο κόσμος ε, εκπαίδευση των μέσων ενημέρωσης. Εγώ θα έλεγα κατάρτιση του ή εκπαίδευση ή καλλιέργεια του κριτικού πνεύματος ε, των μέσων Αυτές είναι οι τροπολογίες 15 και 32. Ένα πιο φιλοσοφικό θέμα. Δεν μου αρέσει ο ρόλος ε, inclusion, χωρίς αποκλεισμούς, που επανέρχεται αναφερόμενος σε ε, στους μετανάστες θα προτιμούσα τον όρο assimilation, ε, ενσωμάτωση και μια φράση ο πολιτισμός ευνοεί την ενσωμάτωση των μεταναστών και άλλων και αυτό βελτιώνει την αρχική διατύπωση που λέει ο πολιτισμός ε, επιτρέπει τον μη αποκλεισμό των μεταναστών, το inclusion. Ε, αυτό ε, δεν αναφέρεται στους μετανάστες που δεν έχουν σκοπό να παραμείνουν σε μια χώρα, αλλά αυτούς που είναι νόμιμοι και επιτρέπεται να παραμείνουν. Υπάρχουν πολλά έργα στο γαλλικό δίκαιο που δείχνουν ότι δεν είναι ε, συνώνυμο. Δηλαδή το inclusion είναι πολύ ελαφρύτερο από το assimilation. Αυτές είναι οι ε, τροπολογίες 15, 18, 23 και 28. Τελευταία ομάδα προτάσεων. Δεν ε, είμαι ένθερμος υποστηρικτής των κατεξουδότηση πράξεων της Κομισιόν, γιατί πολύ συχνά τις ε, βρίσκουν μπροστά μας, και δεν χρειάζονται. Ε, υπάρχουν πολλές στο κείμενο αυτό και βρίσκω κάποιες που δεν είναι απαραίτητες. Υπάρχουν εκτελεστικές πράξεις που αφήνω, αλλά η κατεξουδότηση πράξη είναι οι τροπολογίες 12, 24, 25, είναι περιτές γιατί στην 12 πρόκειται για κατεξοδότηση πράξη που σκοπό έχει τροποποίηση των μη απαραίτητων στοιχείων του παρόντος κανονισμού. Γιατί χρειάζεται να προβλεφθεί αυτό. 24 αφορά την κατεξοδότηση πράξη που εγγυάται την ουσιαστική αξιολόγηση της πρόοδου του προγράμματος. Αυτό δεν αποτελεί θεμελιώδη στόχο και στην 25 είναι οι κατεξοδότηση πράξεις που υπενθυμίζουν το νομικό καθεστώς. Δεν νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίζεται το νομικό καθεστώς κάθε φορά με κατεξοδότηση πράξη. Όλα αυτά είναι περιτά και προτείνω απλά και μόνο την κατάρχησή τους. Κατά τα άλλα, οι πολλές τροπολογίες δεν θα σας κουράσω, είναι, έχουν λιγότερη σημασία, είναι διόρθωση τυπική αλλά όσον αφορά τον πολιτισμό πρέπει να είμαστε ακριβείς. Παραδείγματο χάρη οι 17 και 19 ε, προτείνουν την αντικατάσταση ευρωπαϊκές αξίες με τον όρο αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού γιατί μιλάμε για τον πολιτισμό και πρέπει να μιλάμε για ευρωπαϊκό πολιτισμό εδώ, ε, να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Στην τροπολογία 11 παράδειγμα πάλι προτείνω να, διαγραφεί η μεγαλ, μακροσκελής ε, αναφορά στην Όλαφ. Υπάρχει έτσι κι η Όλαφ. Σε ένα κείμενο που αφορά τον πολιτισμό υπάρχει ρόλος να επιμείνουμε τόσο πολύ στο ρόλο της Όλαφ ακόμα και όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά για τον πολιτισμό καταφέρνει να είναι υπερβολικά γραφειοκρατική. Και Υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που πραγματικά είναι λεπτομερείς και θα, θα σας απαλλάξω. Ελπίζω, ε, αμφιβάλλω αν δεν συμφωνείτε με όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει αυτό το οποίο επιθυμώ είναι να προκαλέσω συζήτηση επ' ενός θέματος που θεωρώ σημαντικό και που αξίζει την προσοχή της Νομικής Επιτροπής. Αξίζει της προσοχής της Νομικής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Ντολβίδη. Ευχαριστώ. Έξοχα κύριε Λεμπρετών παρά είναι καλό το αποτέλεσμα. Δεν ε, κατανοούσα γιατί μας απασχολεί αυτό το θέμα της Επιτροπής δηλαδή νομικών θεμάτων. Εσείς μιλήσατε βεβαίως στην έννοια της προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά ε, ε είναι στην ουσία μία δυνατότητα για να αλλάξει ε, ολόκληρο το κείμενο. Συμφωνώ ότι η ένταξη και το αντίστοιχο ασημιλασιόν δεν είναι το ίδιο πράγμα, στα γαλλικά τουλάχιστον, στα ελληνικά είναι. Νομίζω όμως ότι ασυμιλασιόν δεν είναι όρος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την κοινωνική ένταξη. Για να μην μιλήσουμε για τις αξίες, πώς τις λέτε, πώς τις λέτε, τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μα ακριβώς έτσι αναφέρονται ε, στη χάρτα θέλετε να, ε, να, να δείξετε ότι όλοι είμαστε εναντίον σας αν ε, δεν δεχτούμε τις τροπολογίες σας, μα τα εξέτασα όλα αυτά εκ του ε, όταν μιλάτε αντί για εκπαίδευση και έ την εκπαίδευση για να έχει κανείς κριτικό ε, πνεύμα, αλλά η εκπαίδευση των ΜΜΕ μας δείχνει πώς μπορούμε να πληροφορηθούμε, να μην χειραγωγούμαστε. Δεν νομίζω ότι αυτή η αλλαγή είναι σκόπιμη. Ως προς τη διαγραφή της όλα που επιδιώκεται συχνά, μα θεωρώ ότι δεν μπορούμε να μιλάμε λάβουμε υπόψη την απάτη που έγινε ως προς τα ευρωπαϊκά κονδύλια ή όλα, θα πρέπει να ερευνά για να αποφύγουμε όλες αυτές τις απάτες και καταχρήσεις. Εν πάση περιπτώσει κύριε Λεπρετών άνοιξε η συζήτηση, αλλά δεν πρέπει να σας εκπλήσει το ότι δεν συμφωνούμε. Θα και θα υπάρξει και συνέχεια, γιατί δεν λύγει σήμερα η προθεσμία υποβολή τροπολογιών, έτσι δεν είναι. Oui, le délai pour les... Ναι. Στις 25 Νοεμβρίου λύγει η προθεσμία υποβολής. 27, 27 με συγχωρείτε, λύγει η προθεσμία υποβολή τροπολογιών. Κανένα άλλο δεν ζητάει το λόγο. Άρα τελειώνουμε υπογαλόφωνη σύνθεση. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει την 5 6 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί και θα υπάρχει μια έκτακτη συνάντηση την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου το βράδυ. Δεν ξέρουμε ακριβώς την ώρα, θα την επιβεβαιώσουμε αργότερα. Στο Στρασβούργο βεβαίως. Με αυτές τις ανακοινώσεις σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας σας εύχομαι καλό βράδυ. Γεια σας.